Colleagues, if I could start our... Αρχίζουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Καταρχήν έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για θέματα επιτροπολογίας και ιδιαίτερα των TSI. So, I don't know who we want to δεν ξέρω πώς θα αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε με την Επιτροπή. Ποιος είναι υπεύθυνος από την Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω για ποιο θέμα πρέπει να μιλήσω. Τι περιμένετε από μένα. Μην ανησυχείτε και πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολλοί υπάλληλοι της Επιτροπής δεν ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάνε. Άρα δεν μας εκπλήσει. Και δεν θα έπρεπε να ανησυχείτε γι' αυτό. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί το θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι πολύ περίπλοκο από τεχνικής πλευράς. Καταρχήν, η Επιτροπή Επιτροπή σας εξετάζει ένα προσχέδιο κανονισμού σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα για τηλεματικές εφαρμογές στους επιβάτες. Τα TAP TSI δηλαδή. Under the comitology decision on ε, πρόκειται για μια διαδικασία με έλεγχο. Μπορείτε να αντιταχθείτε αν θεωρείτε ότι έχουμε υπερβεί τις εξουσίες μας ή έχουμε εγκρίνει ε, μέτρα που αντιβαίνουν στο στόχο της Οδηγίας 2008 για τη διαλειτουργικότητα ή εάν αυτό το μέτρο δεν τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τι είναι το TAP TSI είναι μια σειρά προτύπων που έχει καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ε, πολιτές εισιτηρίων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, επεξεργαστούμε τις πληροφορίες, να τις μοιραστούμε εναρμονισμένα σε σχέση με τις ε, τιμές, τους όρους, το, το, πρόγραμμα, τους χρόνους, την, ε, τις αποσκευές και τη μεταφορά τους, την βοήθεια προς τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και άλλες διευθετήσεις όπως μεταφορά δικύκλων στους σιδηροδρόμους και υπάρχουν οι ίδιες εναρμονισμένες ε, πληροφορίες ως προς την πώληση εισιτηρίων και τις πληροφορίες που θα δοθούν στους σιδηροδρόμους, δηλαδή στους σταθμούς σε σχέση με ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Αυτά τα θέματα αφορούν τις διεθνείς ε, μεταφορές. Τα TAP TSI όμως δεν αποτελούν ένα σύστημα ολοκληρωμένης έκδοσης εισιτηρίων για όλο το ταξίδι. Ο ορισμός δεν είναι κωδικοποιημένος και αυτό σας το λέω για λόγους ακριβίας. Μιλάμε για την έκδοση εισιτηρίων, ως προς την έκδοση εισιτηρίων, ένα ενιαίο εισιτήριο, μοναδικό εισιτήριο για μία μετάβαση από το σταθμό μιας χώρας Α στο σταθμό μιας χώρας Β. Ε, με διέλευση από άλλες χώρες, από τρίτη χώρα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ε, επιχειρήσεις. Δηλαδή, έκδοση εισιτηρίων διασυνοριακά. Και ο, η ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίου είναι ένα και μοναδικό εισιτήριο για ένα μόνο ταξίδι χρησιμοποιώντας ε, διατροπικούς τρόπους μεταφοράς, δηλαδή λεωφορείο, μετά τρένο, στη συνέχεια αεροπλάνο και τέλος άλλο ένα λεωφορείο για να φτάσετε από το αεροδρόμιο αύξηση στο τελικό προορισμό. Το TAP TSI λοιπόν δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, αλλά είναι η βάση οικοδόμησης αυτού του συστήματος. Διότι όπως σας είπα, το TAP-TSI είναι ένα κοινό πρότυπο για τη σιδηροδρομική αρχή, τη διαχείριση και την έκδοση εισιτηρίων έτσι ώστε οι επιβάτες που είναι και οι τελικοί ευεργετούμενοι να μπορούν να έχουν κωδικοποιημένες και εναρμονισμένες πληροφορίες. Τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή το TAP TSI, τότε υπάρχουν και επιπρόσθετες εφαρμογές το TAP TSI αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό, καθολικό και ε, διεθνές χρονοδιάγραμμα, ας το πούμε έτσι. Εάν όμως ε, πρόκειται για ε, πληροφορίες ως προς την τιμολόγηση και κάποιος θέλει να ορίσει ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα μετάβασης και να υπολογίσει το χαμηλότερο ναύλο ή τη γρηγορότερη μετάβαση ή εάν επιθυμεί να κλείσει εισιτήρια, να τα αγοράσει, να τα τυπώσει και να κάνει ειδικέ διευθετήσεις για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, τότε χρειάζονται ε, επιπρόσθετες διευθετήσεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ένα μέρος, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, βρίσκεται, εντάσσεται στο TAP TSI. Τα υπόλοιπα, όμως, η έκδοση εισιτηρίων και οι ειδικέ ε, διευθετήσεις για παράδειγμα ως προς την μεταφορά δικύκλων, να έρχεται και ο κύριος Κράμερ, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, όλα αυτά αποτελούν ένα εμπορικό στοιχείο που ίσως αποτελέσει ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των διάφορων ρυθμιστών που ορίζουν την αγορά. Όταν λοιπόν ισχύσουν αυτές οι μεταφορές ε, θα πρέπει να δούμε τη διαχωριστική γραμμή του τι μπορούν να ρυθμίσουν οι δημόσιες επιχειρήσεις και τι αφήνουμε ή αναθέτουμε στην αγορά. Γιατί αυτό αφορά τις επιχειρήσεις πρωτίστως και το θέμα είναι αφορά τις συμφωνίες ΑΙΑΤΑ. Κάποιος μπορούσε να κλείσει μια πτήση Σαμπένα από τις Βρυξέλλες στο Μιλάνο και μετά μια πτήση Αλιτάλια από το Μιλάνο στο Μπάρι. Και να έχει αυτή τη διαδρομή σε ένα ενιαίο χαρτί. Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία ιάτα μεταξύ αεροπορικών γραμμών. Γι' αυτό ε, δεν ίσχυαν οι κανόντες ανταγωνισμού που είχε ορίσει η Κομισιόν. Όμως δεν υπάρχουν πια εισιτήρια επιχάρτου και εάν θέλετε να αγοράσετε ένα εισιτήριο μέχρι το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες Μιλάνο και μετά θέλετε να προχωρήσετε στο μπάρι, να μεταβείτε στο μπάρι, τότε θα πρέπει να κλείσετε ε, σε δύο διαφορετικές ε, στιγμές. Έτσι λοιπόν, Θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή στο όλο αυτό θέμα της τυποποίησης ε, των πληροφοριών και εφαρμογές που είναι δυνατές με βάση τυποποιημένα στοιχεία, τυποποιημένες πληροφορίες ανάμεσα αυτό που μπορεί να ρυθμιστεί από τις, από τις ε, δημόσιες αρχές και τι ε, ανήκει στην αρμοδιότητα του κλάδου. Τώρα βρισκόμαστε στην αρχή της πρώτης φάσης πρέπει να σας πω. διότι η θέσπιση των TAP TSIs μετά από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι το θεμέλιο, το, πρώτο, το θεμέλιος λίθος μιας διαδικασίας που θα ακολουθήσει σε τρεις φάσεις. Έχουμε τη φάση πρώτα του σχεδιασμού του, συστήματος, του ηλεκτρονικού συστήματος, η ανάπτυξή του, και η ε, ε, έναρξη λειτουργίας του. Στα εμπλέκονται πολλοί φορείς, πολλές επιχειρήσεις που φυλάτουν προσεκτικά τα εμπορικά τους μυστικά. Δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν όλα αυτά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες από την εφαρμογή μεγάλων συστημάτων TAP, TAP, TSI για τις, ε, τα εμπορεύματα. Ένα σύστημα που όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, πλειοκτήτες, ε, σιδηροδρομικές, ε, οργανισμοί σιδηροδρόμων κλπ. μπορούν να παρακολουθούν τα, την κίνηση των εμπαρευμάτων. Παρόλο που ο κανονισμός έχει θεσπιστεί πριν από πέντε χρόνια περίπου, υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του συστήματος και θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθούν αυτές οι τρεις φάσεις που ανέφερα, αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει πριν από το 2015. Πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει μέσω ενός φορέα στον οποίο θα συμμετέχουν η Επιτροπή και οι οργανισμοί σιδηροδρόμων, θα εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα ε, πληροφορικής, τα πληροφοριακά συστήματα θα μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό η ταχύτητα της εφαρμογής θα εξαρτηθεί από την προθυμία των ε, εμπλεκομένων φορέων να συνεργαστούν, από τη διαθέσιμότητα ε, κονδυλίων, κονδυλίων στο TSI για το, τα εμπορεύματα. Πήραμε κάποια κονδύλια από τον προϋπολογισμό των TEN-T, των διευρωπαϊκών δικτύων ε, στις μεταφορές. Όλα, όλα αυτά θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το σύστημα που ισχύει για τα εμπορεύματα, όπως σας είπα, το TAF-TSI η Επιτροπή παρόλο που πρόκειται για ένα σύστημα που έχει αποφασιστεί, είναι σημαντικό να καθοδηγήσουμε την όλη διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση. Να αναλάβει, θα αναλάβει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την, τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης που θα πρέπει να ακολουθήσει το σύστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα τμήματα του συστήματος υπάρχουν ήδη με τη μορφή μεμονωμένων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες σε κάποιο βαθμό είναι αρμονισμένες με θελοντικό τρόπο βάσει συστάσεων τα επωνομαζόμενα ε, leaflets, φυλάδια του Διεθνούς Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Δεν μιλάμε εδώ για ένα έργο υποδομής. Δεν κατασκευάζουμε σιδηροδρομικές γραμμές, σταθμούς σιδηροδρόμων ή κάτι άλλο. Απλώς ε, συνδέουμε μεταξύ τους υπολογιστές. Τι θα ακολουθήσει και ολοκληρώνω αυτό. Το TAP TSI, όπως σας είπα, δεν σημαίνει ολοκληρωμένη έκδοση, ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων, αλλά μια έκδοση ενό εισιτηρίου που θα καλύψει μια μακρά διαδρομή που θα περνάει από διάφορε χώρες. Αλλά με, σε συνεργασία με τους ε, σιδηροδρόμους ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε για να περάσουμε στην εφαρμογή του ε, TAP TSI 2, αλλά κάτι που δεν, μπορεί, δεν θα γίνει πριν από το 2016. Το TAP TSI 2 θα διευρύνει τη διαλειτουργικότητα της ενημέρωσης μέσα από τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών στις εθνικές υπηρεσίες. Τα TAP tsi ισχύουν προς το παρόν μόνο για τις διεθνείς υπηρεσίες και θα επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα μεταφορών ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων. Και θα ακολουθήσει και η τυποποίηση ε, διαφόρων εφαρμογών όπως η έκδοση έξυπνων καρτών για, την, ε, για τα εισιτήρια κάτι που υπάρχουν σε επίπεδο εθνικό αλλά δεν υπάρχει τίποτε που να εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα αυτών των συστημάτων μεταξύ κρατών μελών και αυτό είναι ο σκοπός των τεχνικών προδιαγραφών να δημιουργήσουν διαλειτουργικά συστήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Θα ολοκληρώσω λοιπόν λέγοντας ότι το θέμα με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή σας, μάλλον με το οποίο, στο οποίο θα ήθελα εγώ να αναφερθώ, είναι η ρυθμιστική διαδικασία ελέγχου εξέτασης για το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το TAP-TSI και ελπίζω ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις η Επιτροπή σας. Επίσης, έκρινα σκόπιμο να σας μιλήσω για τις μελλοντικές προβλεπόμενες εξελίξεις που θα καταστατούν δυνατές εφόσον εγκριθεί και ξεκινήσει η εφαρμογή του TAP-TSI. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Μα είπε στην αρχή ότι δεν ήξερε το θέμα για το οποίο θα μα μιλήσει, αλλά ήταν μια πληρέστατη παρουσίαση και μα έδωσε λεπτομερή δεδομένα. Και ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να τηρούνται και οι σχετικές νομικές διατάξεις που διέπουν όλο αυτό τον τομέα. Υπάρχει ο κανονισμός του 2007, άρθρο 3.7, και η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του 2008, που επίσης παίζει κάποιο ρόλο. Και το θέμα της ε, τηλεματικής ε, είναι το βασικό θέμα πίσω από αυτές τις ε, τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα και οι δραστηριότητες ε, της Επιτροπής ε, επίσης έχουν αυτό το αντικείμενο και όλες ε, αυτές οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο την τυποποίηση αυτών των προδιαγραφών και γι' αυτό μιλάμε για την έκδοση εισιτηρίων που θα πρέπει να βάλουμε κάποιο στόχο το 2000 15, ε, κάποιο στόχο ε, που βέβαια έχει σχέση και με την απελευθέρωση της αγοράς ε, και τα, οι τεχνικές προδιαγραφές πάντοτε έχουν σχέση με την αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσουν όλα αυτά σε συνδυασμό. Υπάρχει λοιπόν ο τομέας που αναφέρθηκε και υπάρχουν και τεχνικές προδιαγραφές στο τροχαίο υλικό όταν υπάρχουν νέοι μηχανισμοί πέδησης παραδείγματος χάρη ή σηματοδότηση. θα πρέπει να περάσουμε από τις τρεις φάσεις ανάπτυξης. Καταρχήν η ανάπτυξη του σχεδίου, δηλαδή συγκεντρώνονται τα σχέδια που αφορούν ένα συγκεκριμένο ε, υλικό, να δούμε κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα τα δεδομένα, στη συνέχεια εξελίσσεται το σύστημα και στη συνέχεια τίθεται σε εφαρμογή. Έχουμε λοιπόν ε, ένα σύνολο θεμάτων ε, και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει το, Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Μεταφορών, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμο να αναμειχθεί το Κοινοβούλιο στις διάφορες αυτές φάσεις που ανέφερε η Επιτροπή για την όλη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης. Παράλληλα θα πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες πληροφορίες και θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να αναμειχθούν. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν όλα αυτά μας οδηγούν στο στόχο μας, πού υπάρχουν προβλήματα και πού μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τελικά λοιπόν το ερώτημα είναι ε, τι συμβαίνει στα σημεία ε, διασύνδεσης, εκεί που θέλουμε να δουλέψουμε με τρόπο συνδυασμένο. Όχι μόνο ε, δηλαδή να έχουμε πρότυπα για τον σιδηρόδρομο, αλλά όταν έχουμε κάποια σημεία διεπαφής σιδηροδρομικών με οδικές μεταφορές, με πηγαβατικές μεταφορές, με ναυσιπλοεία ή εσωτερική ναυσιπλοεία. Πρέπει να προσέξουμε στα σημεία διεπαφή. Τώρα παίρνουμε απλώς μια πρώτη εικόνα και θα ήταν καλό να μπορούμε να έχουμε αυτά τα δεδομένα πιο συστηματικά για να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία. Γιατί Τώρα απλώς πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες ατάκτως ερημένες και καλό θα ήταν να έχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις τρεις φάσεις της ανάπτυξης και της εφαρμογής και του αρχικού σχεδίου για το τι λογισμικό θα χρησιμοποιείται, αν είναι συμβατό, που υπάρχουν κάποια σημεία που παρεμποδίζεται η διαδικασία, που πρέπει να ανταλλάξουν στοιχεία τα κράτη-μέλη κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Πασκουαρέλη για τις πολύ σαφείς πληροφορίες που μας έδωσε. Ο λόγος που το συζητάμε το θέμα αυτό είναι ότι το θέμα αυτό για την Επιτροπή Μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για τον προϋπολογισμό του 2011 και υπάρχει και ένα πρόγραμμα ε, με τον τίτλο ε, Ευρωπαϊκό Σύστημα Κρατήσεων και Μεταφορών. Ε, δυστυχώς όμως δεν πέρασε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πάντως, η Επιτροπή Μεταφορών θέλει το συντομότερο δυνατόν να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τους σιδηροδρόμους, αλλά στη συνέχεια θα ακολουθήσει και ένα άλλο σύστημα ενιαίας έκδοσης εισιτηρίων για συνδυασμένων μεταφορών. Αυτό είναι ο τρόπο για να κάνουμε τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ περισσότερο ανταγωνιστικέ και περισσότερο ελκυστικέ. Θα του δώσουμε μια νέα ζωή και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Άκουσα ότι πριν από το 2015-2016 δεν πρέπει να αναμένουμε τίποτα συγκεκριμένο και αυτό είναι κάπως απογοητευτικό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Θέλουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων το συντομότερο δυνατόν και το ερώτημα είναι αν έχουμε τα απαραίτητα μέσα, του απαραίτητου πόρους και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι. Δεν μας είπατε σαφώς πόσο θα κοστίσουν όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα είναι μεγάλο το χρηματικό ποσό. Δεν μιλάμε για υποδομή, μιλάμε για τυποποίηση. Δεν ξέρω όμως αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται 5 ή 6 χρόνια για να γίνει. Μιλήσετε και για, τον, για το σώμα που θα έχει τον καθοδηγητικό ρόλο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Τι όργανο θα είναι αυτό. Ο Οργανισμό Σιδηροδρόμων και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα συμμετέχουν από αυτά που έχω ακούσει. Αλλά τι εξουσίες λήψης αποφάσεων θα έχει αυτό το σώμα, πώς, ε, ε, τι σχέσεις θα έχει με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και πώς μπορούν να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις αν ε, θέλουμε να αποκτήσει νέες αρμοδιότητες. Αυτές τις ερωτήσεις ε, ήθελα να σας απευθύνω και κατανοώ ότι προς το παρόν είμαστε πολύ νωρίς, αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε από κάπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάισεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Πασκαρέλη για την πολύ ενδιαφέρουσα εκθεσή του και ευχαριστώ τον κύριο Ελχαντράουι ε, που πήρε να μπει στην ημερήσια διάταξη γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της επιτροπολογίας. Είναι ε, πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητούνται. Και εσείς ε, τονίσατε πολλά σημαντικά θέματα και έχουμε δει και εμείς τη σημασία που έχουν σιδηροδρομικές μεταφορές από την άνοιξη που είχαμε τα προβλήματα με τις αεροπορικές μεταφορές λόγω της ηφαιστειακής τάχτης. Είδαμε πόσο σημαντικές είναι οι εναλλακτικές οδοί μεταφορών. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και διασυνδεδεμένο ακόμη καλύτερα σίγουρα να ξεκινήσουμε από τους σιδηροδρόμους, ε, γιατί ίσως πολλές φορές υπάρχουν στις αεροπορικές μεταφορές τέτοιες δυνατότητες συνδυασμένων εισιτηρίων, αλλά όχι στις σιδηροδρομικές μεταφορές και το Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ νομίζω ότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης ε, πρέπει να συμμετάσχουν και ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών νομίζω ότι πρέπει ε, να συμμετάσχουμε γιατί σαφώς ε, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να βελτιωθεί το σύστημα και η ανταλλαγή δεδομένων είναι σημαντική και πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για την ανταλλαγή δεδομένων. Πρέπει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά τα δεδομένα και αν υπάρχει κάτι για το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά. Σας ευχαριστώ κατευθύν και περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πασκουαρέλη που μίλησε και για τη μεταφορά ποδηλάτων με το σιδηρόδρομο. Είναι κάτι ε, το οποίο διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σε μερικά κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα, σε άλλα όχι και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το προωθήσουμε. Αποφασίσαμε το τρίτο πακέτο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και ε, ε, πολλοί έρχονται και μου λένε ότι στις αεροπορικές μεταφορές δεν υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα γιατί ανεξάρτητα από τις αεροπορικές εταιρείες ε, μπορούν, ε, μπορεί να γίνεται ε, ανταλλαγή δεδομένων ενώ στις σιδηροδρομικές μεταφορές ο κάθε φορέας, η κάθε εταιρεία έχει τα δικά της στοιχεία και νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρξει κάποια ανταλλαγή πληροφοριών και υπάρχει και το τρίτο πακέτο των σιδηροδρόμων που ε, ε, ε, έχει σχέση με αυτό το θέμα. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πληροφοριών. Το συζητήσαμε και το πρωί το θέμα αυτό. Στην Ιταλία είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοση εισιτηρίων διασυνοριακά και εδώ πρέπει η Επιτροπή να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, λαμβάνοντας κάποια μέτρα. Και ένα περαιτέρω βήμα που είναι πολύ σημαντικό είναι το ε, να έχουμε συνδυασμένε ιδιοδρομικέ μεταφορέ. Γιατί η Ελβετία μπορεί να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί πρέπει να περιμένουμε έξι χρόνια μέχρι το 2016 για να εφαρμόσουμε ένα σύστημα που δεν είναι τίποτα καινούριο, δεν πρόκειται για καμιά εφεύρεση, άλλοι το κάνουν ήδη. Και ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα των ε, εμποδίων που μπορούν να υπάρχουν εγώ στο Βερολίνο έχω, την, έχω συνηθίσει να έχω ε, σαφώς ε, την εικόνα του ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσω, με τι δρομολόγια κλπ. Ε, νομίζω ότι εμείς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να φροντίσουμε να προσφέρουμε στους πολίτες της Ευρώπης αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Κράμερ, δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στον κύριο Πασκαρέλη για να ακούσουμε την απάντησή του. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους όσους πήραν το λόγο για να σχολιάσουν ή να διατυπώσουν ερωτήματα. Κύριε Χεράουη, ο κύριος Χεράουι αναφέρθηκε σε κάτι που θα έπρεπε να είχα πει στην αρχή της παρέμβασής μου. Γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, την ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σύγκριση με άλλα μεταφορικά μέσα και πιστεύουμε ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών της πληροφορικής θα μας επιτρέψει να διευκολύνουμε ε, ορισμένες διαδικασίες, ε, κάτι που δεν υπήρχε την παλιά εποχή όταν γράφαμε τα, συμπληρώναμε τα εισιτήρια με το χέρι. Μπορεί να γινόταν, να αρκούσε αυτό να γίνει αν έπρεπε κάποιος να μεταφερθεί από ένα μικρό χωριό στη χώρα Α, σε ένα άλλο μικρό χωριό στην ίδια χώρα ή σε μια γειτονική χώρα. Αλλά τώρα με την εξάπλωση των μεταφορών, κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον ε, χρήσιμο ή ε, αποτελεσματικό. Εκτός από την οδηγία για τη διαλειτουργικότητα υπάρχει και κανονισμός για τους επιβάτες. Υπάρχει λοιπόν μια υποχρέωση για τους οργανισμούς ε, σιδηροδρόμων να προσαρμόσουν τα συστήματα πληροφορικής τους το TAP-TSI και να τα χρησιμοποιούν για την παροχή πληροφοριών και την πώληση και την έκδοση εισιτηρίων. Το TAP-TSI, έτσι όπως ε, ε, ε, υπάρχει αυτή όπως εμφανίζεται τώρα, έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση στο πλαίσιο του, δυνάμει του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί από, με μία γέφυρα ανάμεσα στο TAP TSI και τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Και αυτό είναι ο κανονισμός που ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες της Επιτροπής, που θα δημιουργήσει αυτή τη γέφυρα, αυτό το σύνδεσμο, λαμβάνοντας υπόψη το είδος ε, των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί και εκείνοι που εκδίδουν εισιτήρια με βάση τα αναρμονισμένα ε, πρότυπα του TAP-TSI. Αυτά τα δύο θα κινηθούν ε, σε μια πρώτη φάση παράλληλα. Ο κύριος Καντράου, η κυρία Μάισνερ αναφέρθηκαν στη διακυβέρνηση και στη χρονική συγκυρία για τη διακυβέρνηση είχαμε ε, τη δυσάρεστη εμπειρία της τηλεματικής εφαρμογής στη μεταφορά εμπορευμάτων. Το taf ένα αρμονισμένο σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα σιδηροδρομικά βαγόνια που μεταφέρουν φορτίο. Θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κανονισμό που ζητούσε από τους εμπλεκόμενους φορείς να ε, ε, να φτιάξουν, να εκπονήσουν ένα ε, σχέδιο πανευρωπαϊκό το οποίο καταρτίστηκε με κάποιες δυσκολίες διότι ορισμένοι οργανισμοί σιδηροδρόμων που είναι πιο προχωρημένοι από άλλους στη χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής δεν ήθελαν να ανακαλύψουν τα μυστικά τους που είναι κάτι το νόμιμο αλλά ούτε και την τεχνογνωσία τους να τη μοιραστούν με άλλους τελικά τα καταφέραμε αλλά τώρα που έχουμε πλέον αυτό το στρατηγικό ε, ε, ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει τώρα να εφαρμοστεί διότι υπάρχει αντίδραση, έντονη αντίδραση από πλευράς εμπλεκομένων φορέων να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο με έναν από κοινού και αναρμονισμένο τρόπο. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διακυβέρνηση, η δομή διακυβέρνησης της εφαρμογής είναι αδύναμη και εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση των διαφόρων σιδηροδρομικών οργανισμών. Έστω και αν τεθεί υπό την προεδρία ενός πρώην ε, διευθύνοντος συμβούλου μιας, ε, ενός μεγάλου ε, ε, σημαντικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού οργανισμού αυτό δεν αρκεί και διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πιο ενεργά παρούσα έστω και αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να αφαιθεί στον κλάδο. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια δομή διακυβέρνησης για την υλοποίηση του TAFTSI με μια κοινή Προεδρία από εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο από έναν οργανισμό σιδηροδρόμων. Και αυτή η δομή διακυβέρνησης δεν είναι κάτι που αφορά τις κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη, τις κρατικές αρχές να το αποφασίσουν. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί από τους ίδιους τους χρήστες του συστήματος. Εντοπίσαμε ως μέλη αυτής της δομής διακυβέρνησης την ε, κοινότητα ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, τους διαχειριστές ε, υποδομών, το UITP που είναι η Παγκόσμια Ένωση ε, Μεταφορών, της ενώσεις επιβατών, τους, τις συνδέσμους, τους συνδέσμους πολιτών εκδοτών εισιτηρίων και έχουμε και την τεχνική ε, υποστήριξη που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Αυτό είναι λοιπόν το σχήμα διακυβέρνησης το οποίο έχουμε καταλήξει και στο οποίο πρέπει να παρέμβουμε και εμείς αναλαμβάνοντας ενεργά την Προεδρία του γιατί θέλουμε να ε, προχωρήσει το όλο θέμα. Χρονική συγκυρία. Όπως είπα, η εμπειρία του ΤΑΦ ε, TSA, ήταν απογοητευτική σε επίπεδο διακυβέρνησης και λόγω του ιδιαί... του, της δυσκολίας που προέκυψε όταν χρειάστηκε να ε, συνδέσουμε τα συστήματα πληροφορικής των ε, οργανισμών σιδηροδρόμων που υπάρχουν ήδη, βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τους ειδικού της πληροφορικής. Πρέπει να δεχθώ αυτό που μου λένε ότι θα πετηθεί πάρα πολύ χρόνος. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες σας. Θέλει να προχωρήσουμε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Αλλά είμαι υποχρεωμένο να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή του TAF TSI είναι τρία ή τέσσερα χρόνια. Μάλλον τέσσερα-πέντε χρόνια, όχι νωρίτερα. Από το 2011 γιατί τελειώνει το 2010 μέχρι τις αρχές του 2016, τέλη του 2015. Εγώ και ο διάδοχός μου και εκείνος που θα με διαδεχθεί θα πιέζουμε εκείνους που έχουν αναλάβει την εφαρμογή για ταχύτερους ρυθμούς. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα απόλυτα τα αυτά που μας είπε ο κύριος Κράμερ. Κάτι που όμως νομίζω ότι κατάλαβα είναι ότι μας είπε ότι αυτά τα συστήματα υπάρχουν ήδη και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα ενώσουμε, να τα συνδέσουμε. Δεν, είναι, δεν ισχύει αυτό δυστυχώς. Πράγματι υπάρχουν τα συστήματα, αλλά είναι πιο ανεπτυγμένα σε ορισμένα κράτη-μέλη, πολύ λιγότερο ανεπτυγμένα σε άλλα ή δεν υπάρχουν μάλιστα ε, ή δεν υπάρχουν καθόλου σε άλλα. Ο κύριος Κράμερ έχει την τύχη να προέρχεται από μια χώρα που διαθέτει το καλύτερο σύστημα και γι' αυτό έχει συνηθίσει σε ένα επίπεδο εξυπηρέτησης που οι επιβάτες άλλων χωρών μόνο να τον ηρευτούν μπορούν. Και το να συνδέσουμε αυτά τα διαφορετικά συστήματα που ήδη υπάρχουν και που ήδη λειτουργούν σε βασικά σε εθνικό επίπεδο το γερμανικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ε, κάπως και σε διεθνές επίπεδο. Και κάποιος έκανε τη, έζησε ε, αυτή την εμπειρία πρόσφατα. Αλλά με δυσκολίες. Το να τα συνδέσουμε όλα αυτά, συστήματα που, μπορεί να, που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και δεν, είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει το TAPTSI αλλά πρέπει να δεχθούμε ότι αυτές οι εφαρμογές τηλεματικής είναι, χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αναπτυχθούν. Αλλά ο στόχος που επιδιώκουμε είναι ο ίδιος για όλους μας. Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα με βήμα έως ότου να έχουμε ολοκληρωμένη διαδικασία, διαδικασία, ολοκληρωμένη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων ή ένα εισιτήριο ε, το οποίο θα, θα μπορεί να εκδίδεται σε μια χώρα για, για, να γίνει... για μια διαδρομή που θα καλύπτει πάρα πολλές χώρες, για να γίνουν όλα αυτά θα χρειαστεί χρόνος για να καταλήξουμε σε συστήματα ολοκληρωμένη έκδοσης εισιτηρίων, οπότε τότε ιδιωτικέ εταιρείες, όχι μόνο οργανισμοί σιδηροδρόμων ή πολιτέ εισιτηρίων, αλλά και υπεύθυνοι για την ανάπτυξη λογισμικού θα μπορέσουν να παρέμβουν και να μας δώσουν εφαρμογές τις οποίες θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται μέσω του υπολογιστή του, μέσω του, ενός έξυπνου τηλεφώνου κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Χρειάζουμε την πρώτη βαθμίδα χτίζουμε την πρώτη βαθμίδα του συστήματος αξιοποιώντας πράγματα που υπάρχουν σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης στις ε, χώρες μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πασκαρέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση, αλλά ως προς την Επιτροπολογία, ο κύριος Αλκαντράουι θα ήθελε να επανέλθει. Ναι, ως προς τη χρηματοδότηση δεν έλαβα απάντηση. Ξέρετε ποιο θα είναι το συνολικό κόστος του εγχειρήματος έτσι ώστε να προσαρμόσουμε όλα αυτά τα συστήματα να τα καταστήσουμε διαλειτουργικά και ούτω καθεξής. Και ποιος θα ε, καταβάλει το αντίτιμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ιδιωτικοί φορείς, ιδιωτικοί εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμοστούν. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο επ' αυτού. Και θα ήθελα να προσθέσω και την εξή ερώτηση. Το θέμα χρηματοδότησης είναι το πρόβλημα ουσίας ή περισσότερο τεχνικής υφής ή ένας συνδυασμός των δύο. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν καταβάλουν τίποτα. Μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Αλκαντράουι. Αν απαντήσω ειλικρινά ότι δεν ξέρω, πώς θα σας φανεί θα έχετε δικαίωμα να με πυροβολήσετε. Όχι, δεν θα του επέτρεπα, κύριε Πασκουάλη. Ε, ο πυροβολισμός μπορεί να γίνει μόνο από το Προεδρείο. Μπορώ να σας πω ότι το κόστος είναι περιορισμένο ή σχετίζεται με παράλληλα συστήματα ε, πληροφορικής Έχουμε παράλληλα συστήματα για τα μητρώα, ε, για άδειε οδήγησης, ε, σιδηροδρομικά συστήματα. Έχουμε μια τάξη μεγέθους δηλαδή. Εδώ μιλάμε για την πρώτη φάση της εφαρμογής. της ε, στρατηγικής πρόβλεψης. Η φάση δηλαδή προγραμματισμού με ε, μελέτη αντικτύπου που θα λήξει στα μέσα του 2012. Το TAF-TSI είχε μία μερική χρηματοδότηση από το ten Όμως μόνο ένα εκατομμύριο ευρώ έλαβε από εκεί. Παρά τις δυσκολίες του τάφτου TSI, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ίδια τάξη με γέφους άρα δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης. Είναι ένα πρόβλημα τεχνικής οργάνωσης, όπου αντιστέκονται μερικοί με μονομένη εμπλεκόμενη φορείς. Η χρηματοδότηση όμως δεν είναι το πρόβλημα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Αρχικά μας είπατε ότι δεν ξέρατε, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ξέρατε πολλά και λεπτομερώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος. Η κυρία Σεναλόβα έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Α, μάλλον πριν σας δώσω το λόγο, όταν ε, έχουμε πρώην μέλη που προσέρχονται, τα καλωσορίσουμε. Ο Μάρκ Βότς ήρθε ε, για να συμμετάσχει στις συζητήσεις. Ε, καλωσορίζω λοιπόν, Μάρκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. je obsahově na první pohled převážně technického Eh, zároveň se však eh, jedná o téma, které Νομίζω ότι το θέμα είναι τεχνική υφή, αλλά έχει μεγάλη σημασία και για τις βιομηχανίες και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καταρχήν, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής που σχετίζεται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και οξυδίων του αζότου, καθώς και άλλων μορίων ε, με βάση μικρές, μικρούς σειρμούς, ατμομηχανές, γεωργικά μηχανήματα και ούτω καθεξής. Αυτά τα τρία στάδια θα επαναοριστούν από την 1η Πρώτου 2011, φτάσοντας στο, στο στάδιο 3β. Μιλάμε για τον ε, Ιανουάριο του 2011 και η οδηγία σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν 1.500 ε, επιχειρήσεις. Η οδηγία 2004 κάθετος 26 μιλά για ε, εκπομπές δύο ειδών. Μιλάμε λοιπόν για ευέλικτα συστήματα όπου οι κατασκευαστές θέτουν στην αγορά μηχανήματα που συμμορφώνονται με μηχανές ας πούμε diesel, ατμομηχανές και πλοία για τις πλωτές οδούς ως προς τα οχήματα και τις ατμομηχανές Θεωρούμε ότι παρά το γεγονός ότι μερικοί, μερικοί κατασκευαστές συμμορφούνται με το στάδιο 3β, δεν θα μπορέσουν να ε, θέσουν σε εφαρμογή το πλαίσιο για τις ατμομηχανές βάσει του σταδίου 3β όσον αφορά τους κινητήρες diesel. Ε, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτές τις ατμομηχανές που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον με τύπους 3α. Με τύπο 3α, αν ο τύπος 3β δεν είναι διαθέσιμος. Αυτή η οδηγία δεν αφορά τα πλοία για εσωτερικές πλωτές οδούς. Έτσι, οι κατασκευαστές σε κάθε κατηγορία αυτών των κινητήρων μπορούν να θέσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό που να μην υπερβαίνει το 20% και να σχετίζεται με τις αρχικές εκπομπές. Επίσης, οι μικρές επιχειρήσεις με χαμηλότερο όγκο παραγωγής μπορούν να ορίσουν το ίδιο Όλα αυτά έχουν ε, σχέση με την οικονομική ε, παρακμή και τη μείωση εισοδημάτων. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα σχέδια. Δεν μπορούν βεβαίως όλοι να συμμορφωθούν με αυτά τα δεδομένα, ιδιαίτερα οι μικροί κατασκευαστές. Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής. Προτείνει η Επιτροπή να αυξήσουμε την ποσοστή αναλογία των κινητήρων και να τις εντάξουμε στο ευέλικτο πλαίσιο. Δηλαδή, σε ένα πλαίσιο 20 με 50% ορίζοντας ένα μέγιστο αριθμό κινητήρων που μπορούν να τεθούν στην αγορά των τύπων του τύπου 3α και 3β. Η Επιτροπή επίσης προτείνει το εξής οι κινητήρες για τις ατμομηχανές ε, που θα χρησιμοποιηθούν να ε, ισχύσουν μέσα στο πλαίσιο του 2013, δηλαδή να λήξει αυτό το καθεστώς στο τέλος του 2013. Τέτοια σχέδια ευελιξίας υπάρχουν και στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Δυστυχώς όμως στη Ρωσία, Κίνα και Λατινική Αμερική δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό οι κατασκευαστές από την Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες χώρες, διότι τα ευέλικτα μέσα, μέτρα δεν είναι αρκετά. Ως προς το περιβάλλον, οι βασικοί ρηπογόνοι παράγοντες που αφορούν την, τους ρήπους στην ατμόσφαιρα αφορούν διεξίδιο του άνθρακα και οξίδια του αζότου. Και τα, οι γεωργικοί ελκυστήρες και όλα τα σχετικά ε, ρηπαίνουν το περιβάλλον. το συνολικό ποσό εκπομπών σε κινητήρες δίζελ όταν αλλάξει σε 50% θα πρέπει να συγκριθεί με την παρούσα κατάσταση που ε, είναι στο 20%. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη περίοδος σταδιακής εφαρμογής. Τα επίπεδα όμως εκπομπών θα παραμείνουν αμετάβλητα έχουμε δει και πιο δραστικές αλλαγές στην αρχή της ε, χιλιετίας στο στάδιο 2. Και έτσι οι εκπομπές ε, ακολούθησαν μία φτύνουσα πορεία. Σε σχέση με την άποψη της Κομισιόν και με βάση τις διαβουλεύσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων και αν λάβουμε υπόψη και το περιβάλλον, Πιστεύω ότι πρόκειται για μία ισορροπημένη πρόταση. Θα πρέπει όμως να μας απασχολήσει ο δίκαιος ανταγωνισμός και, τα, και ο οικολογικός εξοπλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι κατασκευαστές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών αυτό θα θέλαμε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Καταναλωτών να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, αλλά ε, είμαι στη διάθεσή σας για να ε, συζητήσουμε για τροπολογίες ιδιαίτερα από τον τομέα του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε κυρία Σεναλόβα. Ευχαριστώ και τη διερμηνέα που κατάφερε να παρακολουθήσει, ευχαριστώ και τη διερμηνέα που κατάφερε να παρακολουθήσει την ομιλήτρια παρόλο που μιλούσε με φοβερή ταχύτητα. Μπορείτε να πάρετε μια αναπνοή τώρα. Ο κ. Νασίκοβιτς από το ΕΛΚ. Μισό λεπτό μπορείτε να περιμένετε. Δεν έχουμε διερμηνία. Μισό λεπτό. Μην προχωρήσετε. Δεν έχουμε ακόμα διερμηνία. Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα μου λένε. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει μικρό τεχνικό ε, πρόβλημα. Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε στη γλώσσα σας αυτό θα έλεγα ότι είναι σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Μήπως θέλετε να κάνετε άλλη μια προσπάθεια να δούμε τι θα συμβεί. Thank you. <clears throat> Szanowny Panie Przewodniczący, chciałbym wskazać na kilka istotnych aspektów, jakie powinny zostać wyszczególnione w przygotowanej przez sprawozdawczynię. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω και όδηση συζητητή από το ΕΛΚ, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά θέματα που πρέπει να καλυφθούν από την έκθεση αυτή. Μιλάμε για την ευελιξία για κινητήρες και Είμαστε ικανοποιημένοι για την τροποποίηση της οδηγίας από την Επιτροπή. Το κύριο πρόβλημα όμως είναι η χρονική καθυστέρηση διότι υπάρχουν δυσκολίες για τους κατασκευαστές που πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε πρέπει να υπάρξουν νέα πρότυπα, θα γίνει η μετάβαση από το 3α στο 3β και αντί να αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο, θα αρχίσει η εφαρμογή το Δεκέμβριο. Ε, δεν πρόκειται εγώ να επαναλάβω όλα τα τεχνικά στοιχεία που μας ανέφερε η συγγήτρια, γιατί είναι υπερβολικά τεχνικά. Εγώ μιλώ απλώς για τα προβλήματα των κατασκευαστών. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και η παραγωγή κινητήρων συνεχίζεται. Πέρυσι είδαμε τα αποτελέσματα της κρίσης. Μειώθηκε η παραγωγή κινητήρων 5-10% και αυτή η μείωση είναι πολύ σημαντική. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούν να διατίθεται σε εμπορία οι κινητήρες παλαιότερης γενιάς, αλλά θα είναι πολύ υψηλότερο το κόστος για τη θέση σε εμπορία και αυτό θα δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλούς κατασκευαστές. Πολλοί κατασκευαστές θα έχουν ζημία. Και ως εκ τούτου θα προσπαθήσουν να κάνουν τη μετάβαση στα νέα πρότυπα για να περιορίσουν τη ζημία που υφίστανται. Είναι μεγάλο το φάσμα των μηχανημάτων που παράγονται και τίθεται σε εμπορία και τα νέα πρότυπα θα τεθούν σε εφαρμογή για όλα αυτά τα μηχανήματα. Επιπλέον, θα είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις εκπομπές, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και βέβαια να μην ξεχνάμε την ασφάλεια. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολλοί κατασκευαστές δεν θα μπορούν να πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα. Πολλοί κατασκευαστές μηχανημάτων δεν, παρά, δεν κατασκευάζουν μόνοι τους ολόκληρο το μηχάνημα, αλλά εξαρτώνται και από άλλους προμηθευτές για εξαρτήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια πρότυπα εφαρμόζουν και φοβούμαι ότι μπορεί να εισάγουμε μηχανήματα που δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την παρουσίαση της ε, εισηγήσής της. Καταρχήν, θέλω να πω ότι εδώ και ένα χρόνο που είμαι στο Κοινοβούλιο πάντοτε ενθουσιάζομαι όταν βλέπω ότι έχουμε μία ε, υποβολή έκθεσης για την οποία δεν έχουμε ε, την έκθεση της ε, καθήλυνα αρμόδιας επιτροπής. Απλώς μια παρατήρηση, είναι μια καινούρια βουλευτού στο Κοινοβούλιο. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τα τεχνικά θέματα. Η κυρία Σανιαλόβα ήδη μας ανέφερε πολλά τεχνικά στοιχεία. Θέλουμε να έχουμε εν γέννη ένα σύστημα το οποίο θα είναι και για το περιβάλλον θετικό και μας ενδιαφέρουν οι εκπομπές από, τα, από τους κινητήρες και όσον αφορά ε, το μονοξίδιο αλλά και τα ε, οξίδια ε, του αζότου και τους υδρογονάνθρακες και τα σωματίδια. Θέλουμε να έχουμε μεταφορές πιο φιλικές προς το περιβάλλον και κινητήρες πιο φιλικούς προς το περιβάλλον. Γι' αυτό προτείνεται από την Επιτροπή μια τροποποίηση της οδηγίας και εγώ θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η τροποποίηση αρκεί να είναι και εφικτή οι προτινόμενες τιμές που προτείνονται ως κατόφλια θα πρέπει να είναι εφικτές και αν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο το αρχικό πρόγραμμα, είναι λογικό να δώσουμε μια παράταση. Αυτό κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θεωρώ σωστό. Και είναι σημαντικό στην ευελιξία την οποία δίνουμε τώρα, δηλαδή περισσότερες συσκευές, περισσότερα μηχανήματα, τα οποία θα μπορούν να τεθούν ε, σε εμπορία κατά τη μεταβατική περίοδο. Ε, είναι ένα μέτρο που ε, πιστεύω ότι είναι σωστό γιατί το ποσοστό που αναφέρεται είναι σωστό, το 20% μπορεί να γίνει 50% μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας και το 0,3% που είναι η αύξηση εκπομπών είναι περιορισμένο ποσοστό. Άρα νομίζω ότι ε, μπορούμε να επιτρέψουμε αυτήν την αύξηση, που είναι τόσο, αύξηση των εκπομπών που είναι τόσο μικρή. Το σημειώνουμε λοιπόν, δεν αγνοούμε τα στοιχεία, αλλά το σημειώνουμε και το παρακολουθούμε. Ε, και για τις μικρές επιχειρήσεις ε, δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο αριθμό, όχι ως ποσοστό των μηχανημάτων που παράγουν, αλλά ως απόλυτο αριθμό και πιστεύω ότι είναι σωστό να δίνουμε αυτή την ευελιξία και για τους μεγάλους και για τους μικρότερους κατασκευαστές και όχι, για όλα τα μηχανήματα, όχι μόνο για τους ε, γεωργικούς ελκυστές, για, τα μηχανή, για τους κινητήρες στη γεωργία και στη δασοκομεία, αλλά και στους σιδηροδρόμους. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ευελιξίας και για, τις, για τους κινητήρες σιδηροδρόμων. Κρίμα που δεν είναι εδώ ο κύριος Κράμερ, που είναι τόσο πολύ φίλος των σιδηροδρόμων και θα χαιρόταν ιδιαίτερα για αυτή την ε, τοποθέτησή μου. Και πρέπει να δούμε ε, μήπως χρειάζεται ένας μετα μια μεταβατική περίοδος ε, για να μην ε, φύγεται και ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών από την εφαρμογή αυτού του μέτρου ευελιξίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λογική η πρόταση της Επιτροπής. Χρειαζόμαστε την ευελιξία. Θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους σε ε, μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την Επιτροπή ο κύριος Βόλγκα. Ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή παρουσίαση αυτής της σύνθετης πρότασης και ίσως πρέπει να επιμείνω στα σημεία που υπογραμμίστηκαν εδώ, στην έκθεση της κυρίας Σναλόβα. Πιστεύω ότι υπογραμμίστηκε η σημασία αυτού του μέτρου για να υποστηριχθεί ο τομέας, ο κλάδος που βρίσκεται ακόμα σε περίοδο μεγάλης κρίσης. Η κατασκευή, οι κατασκευαστές μηχανών ή γεωργικών μηχανημάτων ε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και χρειάζονται κάποια μέτρα στήριξης. Αυτή τη στιγμή όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα μηχανήματά τους θα συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν για τον περιορισμό των εκπομπών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ορισμένες εταιρείες κινούνται προς το στόχο αυτό με μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά πολλές μικρότερες εταιρείες χρειάζεται να ανασχεδιάσουν τα μηχανήματά τους για να παράγουν πιο ισχυρούς κινητήρες, κάτι που έχουν αναλάβει πρόσφατα. Επίσης έγινε αναφορά στις διαδικασίες επιτήρησης με τα κράτη-μέλη θέλουμε να ενισχύσουμε τις διαδικασίες επιτήρησης Υπάρχει τώρα ένα νέο πλαίσιο για την ε, βελτίωση της επιτήρησης ε, της επίβλεψης της αγοράς κάτι το οποίο προσπαθούμε να βελτιώσουμε με τα κράτη-μέλη, ώστε όλες οι, τα μηχανήματα που διοχετεύονται στην αγορά ε, ανταποκρίνονται στα νέα πρότυπα, στους νέους κανόνες. με σκοπό είναι διότι πρέπει, είναι σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος να κυκλοφορούν πλέον μηχαν, κινητήρες και μηχανήματα τα οποία τηρούν αυτούς τους σημαντικούς κανόνες. Ε, χρειάστηκε χρόνος για την προετοιμασία. Ο κλάδος στον Επίτροπο είπε στον Επίτροπο ότι είχε σοβαρές δυσκολίες να, να ανταποκριθεί ε, στα... στους νέους κανόνες για τα επίπεδα εκπομπών. Ανταποκριθήκαμε σε αυτό διατυπώνοντας ε, κάποιες νέες προτάσεις και τελικά εγκρίναμε την πρόταση κειμένου το καλοκαίρι αυτού του χρόνου εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ε, αυτό το κείμενο, ότι το χρειαζόμαστε και το χρονικά περιθώρια ε, προβλέπουν μια καταληκτική ημερομηνία, κάτι που θεωρήσαμε σημαντικό για να δείξουμε ότι δεν υποβαθμίζουμε τα πρότυπα για τις εκπομπές που θεσπίστηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από έξι χρόνια περίπου. Θέλουμε να τηρήσουμε αυτά τα πρότυπα, ε, ε, ε, διατηρώντας όμως κάποια ευελιξία για τα επόμενα τρία χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Κούρνικ. Θέλετε κάτι σύντομα να πείτε. Ο κύριος Κούν. Άλλη μια φορά ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Έχουμε μια παρόμοια κατάσταση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τις οριακές τιμές και για το διοξίδιο του άνθρακος και για τα οξύδια του αζότου, για τα μικρά επαγγελματικά οχήματα. Έχουμε αναφέρει κάποιους στόχους ε, και έχουν εφαρμοστεί και πολλοί από τους στόχους αυτούς και ε, τώρα θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι, ποιος είναι ο στόχος. Εδώ μιλάμε για τη φάση 3α, 3β. Θα είναι διαφορετική η για αυτούς τους κινητήρες από ότι για τα επαγγελματικά οχήματα και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να επιτύχουμε το, το 3β, τη φάση 3β, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ε, προς τα που κινούμεθα. Διαφορετικά κινούμεθα στο σκοτάδι. Ποια είναι τα όρια το σενάριο είναι διαφορετικό σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ε, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μιλάμε για κινητήρες και οι κινητήρες διοχετεύονται στην αγορά, τοποθετούνται σε μηχανές ε, ε, για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετική κατανάλωση καυσίμου, με διαφορετικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν εξετάζουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ούτε την ενεργειακή απόδοση. Αυτή είναι μια συζήτηση, η οποία, αυτό είναι ένα θέμα που αξιολογείται για να βελτιώσουμε την απόδοση αυτών των μηχανών και για να βοηθήσουμε τους χρήστες να ωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν πλέον και που εξελίσσονται σε αυτή την αγορά αυτό που, στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας είναι ε, τρόποι να συμβάλλουμε ε, στην καταπολέμηση της ρήπανσης, της ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε ό,τι αφορά τα νόξ, τα διοξίδια του, του αζότου και τα μικροσωματίδια. Έχουν τεθεί στόχοι. Όταν μιλάμε για το στάδιο 3β, 3α, έχουμε στην οδηγία προσδιορίσει διάφορες κατηγορίες κινητήρων με οριακές τιμές, καθώς και οριακές τιμές. Όλα αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας και αυτή τη στιγμή για τα μικροσωματίδια, αν δούμε τις διάφορες κατηγορίες κινητήρων 130 έως 160 κιλοβάτ, μιλάμε για 0,2 γραμμάρια ανά κιλοβατόρα. 3α, ένα δέκατο. Έχουμε, έχω, έχουμε κατέβει στο ένα δέκατο του 3β. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος με αποτέλεσμα να μπορέσουν να περιορίσουν τις εκπομπές τους τα κράτη-μέλη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, πολύ. Θέλει κάτι να μας πει η συγγήτρια, υπομορφή ε, συμπεράσματο. Όχι, δεν έχω κανένα σχόλιο. Εντάξει. Προβλέπουμε τη 16η Νοεμβρίου για προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Στις 25 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και ως προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν ξέρουμε τι προτίθενται να κάνουν ο συνήθως και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Ολομέλεια. Εμείς όμως έχουμε τη 16η ε, Νοεμβρίου για υποβολή τροπολιών και στις 25 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή. Θα διακόψουμε για μισή ώρα πριν συζητήσουμε με τον κύριο Γκουντούλ από την ΕΑΣΑ. Άρα θα επανέλθουμε στις 5 παρατέταρτο για να συζητήσουμε με τον κύριο Γκούντου. Okay, colleagues. Can we Συνάδελφοι. restart the meeting? We have. η συνεδρίασή μας. Έχουμε τον κύριο Γκούντου από την ΑΙΑΣΕ, τον ε, ΑΙΑΣΕ, τον εκτελεστικό διευθυντή της ΑΙΑΣΕ για αυτή τη συζήτηση Είχαμε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέματα που απασχολούσαν τα μέλη μας και σκοπός μου είναι να δώσω το λόγο στον κύριο Γκούντου αρχικά και μετά θα διατυπώσουμε ερωτήσεις και θα κάνουμε σχόλια. Κύριε Γκούντου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να εμφανιστώ ακόμα μια φορά στην Επιτροπή Μεταφορών. Είμαι ευτυχής γιατί ακόμα μια φορά μπορώ να έχω μαζί σας ε, με τα μέλη της Επιτροπής σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την ε, αμέριστη υποστήριξη που έδωσε στην ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας και προτίθεμαι να σας δώσω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ε, που θέλετε να αποκτήσετε για τον οργανισμό. Θα πω δύο λόγια για τη γενική κατάσταση του οργανισμού και θα σας μιλήσω για τη στρατηγική μας σε θέματα ασφάλειας ε, τις αεροπορίες, εφόσον αυτό είναι το αντικείμενό μας, το θέμα μας, από τη θέσπιση το Νοέμβριο του 2009 της τροπολογίας 1108 στο βασικό κανονισμό 2016 2008 ο οργανισμός είναι αρμόδιος για την σύνολο της ασφάλειας ε, των πτήσεων ε, σε όλα τα επίπεδα, από την αυσιπλοεία μέχρι τα αεροδρόμια. Φέτος έλαβε ενεργά μέρος ο οργανισμός στην προετοιμασία και στο συντονισμό μάλιστα των ε, ε, ευρωπαϊκών φακέλων που με επιτυχία υποβλήθηκαν στην ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου και στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου του ΙΚΑΟ στην οποία στη Γενική Συνέλευση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο η Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τη δημιουργία πριν από ένα χρόνο μιας ομάδας εργασίας European Aviation Safety Advisory Committee με, που προεδρεύεται από τον οργανισμό από την ε, ΕΑΣΑ τον Ευρω... το τον κλάδο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια κράτη-μέλη. Η ομάδα αυτή έχει αναλάβει να παρέχει συμβουλές σε θέματα ασφάλειας πτήσεων, να περιγράφει το πρόγραμμα για την ασφάλεια της αεροπορίας το ευρωπαϊκό και να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια της αεροπορίας στην Ευρώπη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΚΑΟ το πρόγραμμα, είναι το πρώτο πρόγραμμα δράση και το πενταετέ πρόγραμμα δράση υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το Δεκέμβριο αυτού του έτου, και ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά μια έγκριση στο ανώτατο ε, ποιολητικό επίπεδο αυτού του σχεδίου δράση θα αποτελέσει μια ουσιαστική βάση για τη βελτίωση τη ασφάλεια αεροπορία στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας το 2009, εφόσον δεν έχουμε ακόμα ε, ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία για το 2010. Η ασφάλεια, τα επίπεδα ασφάλειας ήταν εξαιρετικά το 2009. Είχαμε μόνο ένα ατύχημα στον τομέα της εμπορικής ε, αεροπορίας και δύο θανατηφόρα ατυχήματα, θανατηφόρα ατυχήματα στην εμπορική αεροπορία με ελικόπτερο που είναι πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά στατιστικά στοιχεία. Τα χαμηλότερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι συστάσεις που ε, υποβάλλονται από τους ερευνητές των ατυχημάτων διπλασιάστηκαν από το 2008 μέχρι το 2009 με διεύρυνση των αρμοδιοτήτων σε άλλους τομείς της αεροπορίας. Αυτή η τάση θα οπωσδήποτε θα αυξηθεί, δημιουργώντας έτσι ένα πρόσθετο, σημαντικό πρόσθετο <clears throat> φόρτο εργασίας <clears throat> για τον οργανισμό. <clears throat> Σε ό,τι αφορά τι εκθέσεις για τυχήματα που δέχεται ο οργανισμός, αυξάνεται σταθερά. Έχουμε την υποχρέωση να αναλύσουμε αυτά τα ατυχήματα για να αντλήσουμε τα αναγκαία διδάγματα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας. Αυτό μας οδήγησε να, ιδρύσουμε, ε, να δημιουργήσουμε ένα ειδικό εργαλείο που μας επιτρέπει με επαγγελματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό τον αυξημένο φόρτο εργασίας. Τώρα θα σας μιλήσω για την δραστηριότητά μας σε κανονιστικό επίπεδο που υπήρξε σημαντική το 2009 και το 2010, κάτι θα συνεχίσει και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Το 2009 δημοσιεύτηκαν 12 notice of proposed amendments, ειδοποίηση για προτινόμενες τροπολογίες. Δύο πολύ σημαντικά. Το ένα αφορά τη συμβατότητα, την επιχειρησιακή ε, των αεροσκαφών και το δεύτερο τους κανόνες εφαρμογής OPS. το τέλος του 2009 η Επιτροπή μας ζήτησε μια ταχεία διαδικασία, fast track, για να μεταφέρουμε τρεις ισχύοντες κανόνες που αφορούν το Air Traffic Management, το ATM, ώστε να θεσπιστούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας πριν από το τέλος του 2010. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τις άδειε των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τις απαιτήσει για τους ελεγκτές και τις απαιτήσει για τις αρχές ε, που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση της ε, αεροπορίας υποβάλαμε στην Επιτροπή τις προτάσεις μας το Μάρτιο με εμπρόθεσμα αυτοί οι τρεις κανονισμοί που απλώς μεταφέρουν, ενσωματώνουν τους ισχύοντες κανονισμούς θα εξεταστούν περαιτέρου ώστε να εντάξουν όλα τα στοιχεία και όλες τις απαιτήσεις του βασικού κανονισμού. Το 2010 Έχουμε, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο υποχρεώσεων. Θα ε, εξετάσουμε τα σχόλια για το ΟΠΣ, τις απαιτήσει για τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές, τις γνωμοδοτήσεις του οργανισμού για το FCL και το ιατρικό σκέλος. Η ομάδα εργασίας MDM 055 διατύπωσε, διατύπωσε προτάσεις για τους περιορισμούς του, του, του χρόνου πτήσης, FTL, Flight Time Limitation. Θα επανέλθω λεπτομερώς μετά από τις ερωτήσεις σε όλα αυτά τα σημεία. Η προτεραιότητα που δίνουμε στην επεξεργασία νέων κανόνων για, που θα καλύψουν τις νέες αρμοδιότητες δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις, ε, παρα, τις διατάξεις του κανονισμού για την airworthiness. Για το μέλλον θα ήθελα να σας μιλήσω για τη θαυμάσια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον Eurocontrol που έχει δημιουργήσει μια ειδική διεύθυνση. Ε, υπάρχει και ένα γραφείο σύνδεσμος με τα θεσμικά όργανα στο Eurocontrol που υποδέχεται εκπροσώπους του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τους εμπειρογνώμονες του Eurocontrol που θα εργαστούν υπό τον, την εποπτεία του ε, για τη, σε θέματα τυποποίησης ATM, αναλύσεις ασφάλειας ATM κλπ. Εξάλλου, μια ανταλλαγή εκπροσώπων μεταξύ PRP και ΛΕΑΣΑΚ εγγυάται ότι οι στόχοι ασφάλειας ATM θα οριστούν με ακρίβεια και θα τηρούνται με αυστηρότητα. Τώρα θα ήθελα να ασχοληθούμε με το χρηματοδοτικό. Ο προϋπολογισμός του 2010 ανέρχεται σε 107 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατομμύρια προέρχονται από τη βιομηχανία ε, με βάση τα έσοδα και το υπόλοιπο αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πέρα από τα 107 εκατομμύρια υπάρχει ένα αποθεματικό, ένα πλεόνασμα που ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες το 2010 έχουν ως εξή. Τίτλος 1 προσωπικό 56 εκατομμύρια, Τίτλος 2 Διοικητικές δαπάνες 14 εκατομμύρια ευρώ. Τίτλος, τίτλοι 3 και 4 Λειτουργικές δαπάνες 40 εκατομμύρια ευρώ. Στα πλαίσια των 40 εκατομμυρίων τα 25 αφορούν τις υποβολαβίες που αναθέτουν οι εθνικές αρχές. έχουμε 570 προσωρινούς και περίπου 520 θα, θα ανέλθουν σε 520 στο τέλος του έτους. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και 55 συμβασιούχους. Για το 2011 δεν θα αλλάξει άρδινο προϋπολογισμός. Το business plan, το πενταετές προβλέπει 37 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση όμως την χρηματοπιστωτική κρίση, η Επιτροπή προβλέπει η ευρωπαϊκή εισφορά να παραμείνει, να μειωθεί κατά 3 εκατομμύρια σε σχέση με το προγενέστερο business plan. Βεβαίως αυτό δεν είναι ευπρόσδεκτο τη στιγμή που οι αποστολές είναι περισσότερες και οι δραστηριότητες επίσης η βοήθεια από το Eurocontrol για το ATM είναι ευπρόσδεκτη. Ως προς τις προσλήψεις, το πρόγραμμα του 2011 δεν θα διαφέρει. Δηλαδή 514 έναντι 70 συμβασιούχων, άρα δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε για τις μελλοντικές αποστολές. Θα πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό. Ε, ως προς τις εισφορές, θα ήθελα να διορθώσω την αντίληψη που υπάρχει, ότι δηλαδή έχουμε περισσότερους, ε, περισσότερες προσόδους από τις αναγκαίες. Το 2007 το πλεόνασμα που είχε εγγραφεί οφελόταν, οφειλόταν στην αλλαγή μεθόδων πληρωμής. Τον ίδιο χρόνο είχαμε τις πληρωμές για τη λήξη ανάθεσης έργων και τις πληρωμές υπό μορφή προκαταβολής για μελλοντικές εργασίες. Το 2008 και 2009, ιδιαίτερα το 2009, το πλεόνασμα εξαλείφθηκε διότι είχαμε περισσότερα έργα ως προς, τη, προς τα έργα ε, σε σχέση με το παρελθόν. Προτείναμε στην Επιτροπή να τροποποιήσουμε τον υπάρχοντα κανονισμό ως προς τις εισφορές ε, και τους μισθούς, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα για τα πραγματικά έργα και να μπορέσουμε να καταβάλουμε τις αμοιβέ για την ε, ανάθεση, ευρύτερη ανάθεση έργων. Δεν θα υπάρξει μία αύξηση κόστους από τις επιχειρήσεις και ελπίζουμε η Επιτροπή να εγκρίνει αυτό το νέο κανονισμό τάχιστα. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι ο οργανισμός ακολουθεί το ISO 900 9001 και ο εσωτερικός έλεγχος έτυχε διεθνούς πιστοποίησης. Αυτό ε, δείχνει τον επαγγελματισμό του οργανισμού ως προς την ποιότητα και τους ελέγχους. Αυτή είναι η αρχική μου δήλωση και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις και να ε, συμπληρώσω ε, περαιτέρω πληροφορίες, ό,τι άλλο θα θελήσετε να μάθετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τον κύριο Γκουντού. Εντυπωσιακό ο απολογισμό που μας παρουσιάσατε. Όχι μόνο για τον προπολογισμό του 2010, που έχει αυξηθεί και αποτελείται κατά 2 τρίτα από χρηματοδότηση που προέρχεται από τον κλάδο και κατά 1 τρίτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ε, σημαντικά τα καθήκοντα τα οποία ε, αναλαμβάνεται. που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες ε, συζητήσαμε πολλές φορές πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα θέματα ασφάλειας μέσω του ground handling και όσον αφορά τον έλεγχο επιβατών και όπως ε, διδαχθήκαμε προσφάτως τα κενά που εντό εισαγωγικών υπάρχουν στη μεταφορά εμπορευμάτων. Ο τομέας σας περισσότερο στρέφεται γύρω από την τεχνική επαλήθευση και τον τεχνικό έλεγχο των operators ε, των ε, αεροπορικών εταιριών και επίσης είναι σημαντικό να μην υπάρχει κανένα λάθος και αυτό το οποίο συνέβη στην Νοτιοανατολική Ασία με το Α480 και με τον ε, στροβιλοκινητήρα που υπέστη ε, κάποια ζημία και αναγκάστηκε μια αναγκαστική, έγινε απαραίτητη μια αναγκαστική προσγείωση και ποιες είναι οι συνέπειες. Η ασφάλεια των πτήσεων στην Ευρώπη είναι ένα σημαντικό αντικείμενο στα πλαίσια των καθηκόντων σας. Και ο καταμερισμός της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών. Ποια είναι τα σημεία διεπαφής μεταξύ του Βόρειο Ευρωπαϊκού, Κεντρικού Ευρωπαϊκού και Νότιου Ευρωπαϊκού χώρου. Ο απολογισμός ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Μας είπατε ότι το 2009 δεν υπήρχαν ε, ε, ατυχήματα, μόνο το ατύχημα με το ελικόπτερο με δύο θύματα. Και είναι πολύ σημαντικό να ε, τονίσουμε ότι στην Ευρώπη πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές. Και εδώ απαιτεί τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Και στην Επιτροπή Μεταφορών το έχουμε ήδη συζητήσει. Όταν έχουμε ατυχήματα στις αεροπορικές μεταφορές, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την έρευνα και το συντονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Υπάρχει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία στη Γερμανία, υπάρχει η Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που μπορούν να συνδυάσουν τις αρμοδιότητές τους ε, και τους πόρους που διαθέτουν για να βελτιώνονται οι έρευνες και να παράσχουν βοήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων και συνεργατών, είπατε ότι έχει 520 εργαζομένους προσωρινούς θα μπορούσατε να μας πείτε πώς βλέπετε και στο μέλλον την εξέλιξη του προσωπικού, τι είδου συνεργάτες και αναφέρετε ένα προϋπολογισμό 57 εκατομμυρίων. Ε, θα μπορούσατε ίσως να μας αναλύσετε πώς θα καταβάλουν οι αμοιβές του διάφορους συνεργάτες. Πάντως ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την έκθεσή σας. Ο κύριος Ελ Καντραουή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουντού για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τακτικές επαφές και να μας ενημερώνετε για το έργο σας. Έχω σημειώσει κάποιες ερωτήσεις. Ε, καταρχήν, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ασφάλεια και είναι εξαιρετικά τα στοιχεία που μας αναφέρατε για το 2009. Όμως ε, κάποια συμβάντα υπήρξαν πρόσφατα με τους κινητήρες Rolls-Royce, παραδείγματος χάρη. Και μόλις ολοκληρώσαμε το νομοθετικό μας έργο όσον αφορά ε, ε, την ευθύνη για τα ατυχήματα είναι η έκθεση ΒΕΡΑΚ. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το νομοθετικό κείμενο σας ικανοποιεί και ποιος είναι ο δικός σας ρόλος ε, στην έρευνα σε τέτοια συμβάντα, όπως ε, και στην περίπτωση του αεροσκάφους ε, στις Αυστραλιανές αερογραμμές. Ξέρω ότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν αφορά ευρωπαϊκή εταιρεία, όμως είναι ένα αεροσκάφος που κατασκευάζεται στην Ευρώπη και μας ενδιαφέρει. Θα ήθελα τη γνώμη σας λοιπόν γι' αυτό. Αναφέρατε και τους πόρους και είπατε ότι είναι 3 εκατομμύρια λιγότερο προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά θα μπορούσαν και να αλλάξουν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. 3 εκατομμύρια λιγότερο σε σχέση με το επιχειρησιακό σας σχέδιο. Θα δυσκολεύσει τη δουλειά σας αυτό. Και αναφέρεται και νέα καθήκοντα για το μέλλον. Για τα νέα καθήκοντα, σε τι τομεί θα χρειαστείτε επιπλέον προσωπικό, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμη, αναφέρεται νέες διατάξεις όσον αφορά τα τέλη και τις εισφορές. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάποιες αρχές που διέπουν αυτές τις τροποποιήσεις σε σχέση με το τωρινό σύστημα, τι αλλάζει και πώς θα επηρεάσουν οι αλλαγές αυτές τα έσοδά σας. Τέλος, έχω και κάποιες ερωτήσεις που συζητάμε εμείς τους τελευταίους μήνες. Μιλήσατε για το χρόνο, για το περιορισμό του χρόνου πτήσης συμπεριλαμβάνεται και το θέμα του χρόνου ανάπαυσης. Το συζητήσαμε πριν από έξι μήνε ε, και στο μεταξύ νομίζω ότι μια ομάδα εργασία θα έπρεπε να συνεδριάσει και θα έπρεπε να έχει αποτελέσματα μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν μπορείτε, ενημερώστε μα και για το τι ισχύει τώρα. Άλλο ένα παρόμοιο ερώτημα τώρα. για ένα θέμα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και αφορά τις άδειες των κυβερνητών. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας θέση. Ποιες αρχές θα θέλατε εσείς να ισχύσουν. Μια τελευταία ερώτηση τώρα. Στην εισαγωγική σας παρουσίαση μιλήσατε για το Single Sky. Ε, ποια είναι η σχέση με το ΣΕΖΑΡ και ποια είναι η σχέση με τη δουλειά τη δική σας. Ε, πώς συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας στο Single Sky. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκουντού για την παρουσίαση που μας κάνατε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που ήδη άκουσα από τους προλαλήσαντες, αλλά ένα σημείο θα το επαναλάβω, γιατί είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι ο αριθμός των ατυχημάτων μειώθηκε τόσο πολύ και νομίζω ότι είναι πρωτοφανές που έχουμε τόσο χαμηλό αριθμό ατυχημάτων και εύχομαι να παραμείνει τόσο χαμηλός και στο μέλλον. Για την έκθεση Βεϊράκ επίσης θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ασχολείστε και με αυτό το θέμα και θέλουμε να έχουμε Σωστέ έρευνε σε περίπτωση ατυχημάτων. Άκουσα που το ανέφερε και ο κύριο Ελκαντράου και είναι σημαντικό. Τώρα, ε, σε σχέση με την ασφάλεια πτήσης κατά την περίοδο της ε, ηφαιστειακής στάχτης, η ΕΣΑ ε, αναμίχθηκε στην διαδικασία για την διασφάλιση της ασφάλειας. μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι δεν ε, ε, ισχύουν ε, οι πιο αποτελεσματικές λύσεις. Νομίζετε ότι τώρα υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός ώστε στο μέλλον να έχουμε καλύτερη έρευνα, καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερες εγγύσεις για την ασφάλεια. Επίση υπάρχει το θέμα τη τεχνολογία ε, στο θάλαμο διακυβέρνηση του αεροσκάφου, ε, Όλο και περισσότερη τεχνολογία ε, και θα ήθελα να μας πείτε αν νομίζετε ότι στο μέλλον οι πιλότοι θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερες σπουδές για να μπορούν να χειριστούν τα πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα και αν θεωρείτε ότι με τις συσκευές αυτόματου πιλότου ε, μπορούμε να έχουμε καλύτερη πλοήγηση του αεροσκάφους από ότι με τον ε, άνθρωπο ως κυβερνήτη του αεροσκάφους. Έχουμε λάβει και αρκετά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πιλότους που πήραν άδεια στις ΗΠΑ. Πολιτείες ενώ στην Ευρώπη δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρουν ε, τέτοια αντίστοιχη άδεια. Και αυτές οι αμερικανικές άδειες ενδέχεται να ε, επιτραπούν και στην Ευρώπη. Ε, θα επιτραπούν μόνο για, τις, ε, για αμερικανικά αεροσκάφη ή μπορεί να επιτραπούν αυτές οι άδειες και στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες άδειες που είναι ασφαλέστερες από κάποιες άλλες. Μας ενδιαφέρει η εναρμόνιση, αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει η ασφάλεια. Υπάρχει μόνο κάποιος που πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένα μέλος του πληρώματος αεροπλάνου. Ο κύριος Ολύρη, Κύριε Λίντεμπεργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Οι ερωτήσεις για την έκθεση Βεράκ έχουν ήδη γίνει και δεν θα τις επαναλάβω. σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις και μηνύματα που παίρνουμε από διάφορους πιλότους, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας. Ποιος, ποια είναι η αιτιολόγηση για την απόφαση που έχετε λάβει. Αυτό θα θέλω να μας πείτε. Επίσης υπάρχει ο κανονισμός για το code sharing και για το wet leasing. Πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε. Ε, εδώ τίθεται θέμα αεροσκαφών από ε, τρίτες χώρες στο θέμα, στον τομέα του wet leasing και ε, για την εφαρμογή του OPS και των διατάξεων για το πλήρωμα καμπίνας. Είναι θέματα που τα έχουμε συζητήσει και έχουμε μιλήσει ε, για την ανάγκη του να έχουμε διατάξεις για το χρόνο ανάπαυσης και μας ενδιαφέρει να μας πείτε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε το τι έχει γίνει, γιατί και στην ε, προηγούμενη ε, θητεία είχαμε παρακολουθήσει το θέμα. Είμαι και εγώ ένας από τους δεινοσαύρους που ήταν εδώ και την, κατά την προηγούμενη περίοδο και αυτό τα οποία είχαμε συζητήσει τότε δεν θα θέλω να πάνε χαμένα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ε, ε, ποια είναι τα επιχειρησιακά συμπεράσματα στην πράξη από την ε, υπόθεση της ηφαιστειακής τάχτης έχετε καταλήξει στο ότι πρέπει να έχουμε νέα συστήματα, νέες συσκευές μέτρησης, χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες διατάξεις για την ασφάλεια, για την ασφάλεια των δεδομένων. Υπήρχαν ε, κάποια θέματα που δημιούργησαν μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι θα έπρεπε και εδώ υπάρχει και το θέμα της καταστρατήγησης ε, των ε, δικαιωμάτων των επιβατών και προσωπικά δεδομένα των επιβατών τα οποία ε, κοινοποιήθηκαν και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω από εσά ποια είναι τα μέτρα που κατά τη γνώμη σας πρέπει να ληφθούν για να μπορεί να αποτραπεί μια τέτοια κατάσταση στο μέλλον. Δεν θέλω να ξαναζήσουμε μια τέτοια κατάσταση έκρηξης ηφαιστείου, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσε και να ξανασυμβεί. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Γκούντι. Ίσως δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη με τα πράγματα όπως άλλοι συνάδελφοι. Αυτό που αναφέρθηκε είναι τα email τα οποία λαμβάνουμε όχι μόνο από τον κλάδο αλλά και από τους ε, ψηφοφόρους μας, όχι για τον τομέα της εμποριακής αεροπορίας, αλλά μιλάμε για το gliding, ε, για την, ε, τα μικρά αεροσκάφη ψυχαγωγίας. Ε, υπάρχουν, ε, ε, έχουν διατυπωθεί παράπονα. Εμείς είμαστε υπέρ της ίδρυσης της ΕΑΣΑ. Δεν θα αρχίσω να κάνω σχόλια για τους κινητήρες. οι κινητήρες, οι κινητήρες χαλάνε καθημερινά παντού στον κόσμο και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε εδώ. Αλλά πέρα από αυτό αυτό που με προβληματίζει εμένα, μετά από συνομιλίες που είχαμε εκπροσώπους του κλάδου, ποια είναι η εντολή της ΕΑΣΑ. Διότι έχω την εντύπωση ότι υποστηρίξαμε την δημιουργία αυτού του οργανισμού, ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού, για θέματα ασφάλειας, όχι για θέματα περιβάλλοντος ή για θέματα κοινωνικών υποθέσεων. Ο ρόλος σας και η εντολή σας είναι η ασφάλεια καλείστε να ασχολείστε με τα θέματα ασφάλειας. Το κάνετε. Δεν ξέρω τι γίνεται μεταξύ ΆΣΑ και Επιτροπής, αν υπάρχει κάποια σύγχυση μεταξύ των δύο. Βλέπουμε τη διαδικασία ε, σύνταξης κανόνων και κανονισμών. Και έχω την εντύπωση ότι ασχολείστε με πολλά άλλα πράγματα, όχι αποκλειστικά με τα θέματα της ασφάλειας. Βεβαίως υπάρχουν διμερείς ε, συμφωνίες που εξακολουθούν να ισχύουν διότι είναι σύνθετο το θέμα, αλλά οι εξεταστές στο, ε, στην εκπαίδευση στους προσημειωτές ε, έχουμε το πλήρωμα θαλάμου επιβατών χρειάζονται κάθε γίνεται ε, έλεγχος ιατρικός κάθε έξι μήνες. Όχι. Είναι θέμα ασφαλείας, είναι θέμα ασφαλείας η παρουσία πληρώματος στα αεροσκάφη. Δεν είναι ρόλο της ΕΑΣΑ να λέει πόσοι, πόσα πρέπει να είναι τα μέλη του πληρώματος σε ένα αεροσκάφος. Και όλα αυτά τα θέματα ε, καλύπτονται από κάποιο νέφος με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που δεν θα είναι καθόλου ικανοποιητική και το θέμα του περιορισμού του χρόνου πτήσεων. Ζητούν τις απόψεις μας, τους δίνουμε τις απόψεις μας και κανένας δεν μας ακούει. Αλλά αυτό δεν ίσχυε με τον περιορισμό του χρόνου πτήσης. Έκθεση μήμπας είναι κάτι το τελείως παράλογο. Δεν ξέρω ποιος το προώθησε αυτό και όμως ήταν ένα άκρος αμφισβητήσιμο κείμενο αντιλαμβάνομαι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εσάς από το μηδέν να δημιουργήσετε έναν οργανισμό που πρέπει να τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης. Η δουλειά σας θα είναι πάντα, δύσκολη. Δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά πρέπει να ακολουθήσετε, κύριε Γκουντού, τη σωστή κατεύθυνση. Το λέω σε εσά και στα μέλη της Επιτροπής. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να εστιαστείτε στα θέματα της ασφάλειας. Τα άλλα θέματα θα αντιμετωπίζονται αλλού, διότι θέλουμε μια παραγωγική βιομηχανία στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη ε, ε, πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνετε σε θέματα που δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι ο τομέας σας, διότι ε, βλέπουμε να διαμαρτύρονται οι ψηφοφόροι μας και θέλω να, να δείτε, να δείτε, να περιοριστείτε, να περιοριστείτε σε αυτά που υπάγονται απόλυτα στην αρμοδιότητά σας. Διότι αν δεν το κάνετε αυτό, άνθρωποι σαν και εμένα θα εξακολουθούν να διαμαρτύρονται απευθυνόμενοι σε εσά και στα μέλη της Επιτροπής. Θέλουμε ο οργανισμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά, να ε, οι προσπάθειές του να στεφθούν με επιτυχία εφόσον θα περιορίζεται στο τομέα στις αρμοδιότητες οι οποίες του έχουν ανατεθεί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκουντό, δεν... εγώ πρέπει να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε. Δεν... Ε, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το πλήρωμα. Πριν από λίγα χρόνια, εδώ και αλλού, είχαμε συζήτηση, συζήτηση έντονη για τη ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. Όχι μόνο στη διάρκεια μιας μέρας, αλλά είχαμε μιλήσει και για στη διάρκεια μιας εβδομάδας και για διάρκεια 30 ημερών και είχαμε πει κατά πόσο τα διαστήματα αυτά είναι ικανοποιητικά. Δεν θέλω να εμφανίζομαι σαν, σαν ε, ένας δεν θέλω να είμαι σαν ένας γιατρός από τον οποίο ζητήθηκε να δώσει μία γνώμη και είπε ότι αυτή πρέπει να είναι η χρόνια ανάπαυσης. Δεν ζηλεύω αυτά που κάνετε εσείς. Εσείς επιλέξατε αυτό το ρόλο, αλλά πρέπει να υπάρξει ομοιομορφία. Η ομοιομορφία είναι ιδιαίτερα σημαντική εδώ οι άδειες, ε, η χορήγηση αδειών στους πιλότους και οι κανόνες για τη χορήγηση αυτών των αδειών. Πιστεύετε ότι πρέπει να είναι μηχανικοί οι και μηχανικοί ή μόνο πιλότοι πρέπει να είναι... Ε, πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση, ειδική κατάρτιση ε, τι θα κάνουν αν σταματήσει ένα κινητήρα, αν δεν λειτουργεί ο αυτόματος πιλότος, θα είναι σε θέση να προσγειώσουν το αεροσκάφος. Και οι επιστολές που ανταλλάσσουμε με αυτά τα θέματα ασχολούνται. Το, ο ενιαίος ουρανός, το ΣΕΖΑΡ, θα αρχίσει να λειτουργεί το 2015 έχουν γίνει κάποιες ρυθμίσεις για την κεντρική Ευρώπη. Ήμουν στην Τσεχία ο εισηγητής για αυτό το θέμα πριν από 8 περίπου χρόνια. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία υπάρχουν, όπως το Σέζαρ που ε, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται προοδευτικά και σκέφτομαι τα μεγάλα αεροσκάφη Κάποιοι από τους εμπειρογνώμονές σας αισθάνονται ότι αυτά τα μεγάλα αεροσκάφη είναι ασφαλή. Μειώσατε και σας συγχαίρω γι' αυτό τα ποσοστά ατυχημάτων. Δεν έχουμε ακούσει για ατύχημα για ενός μεγάλου αεροσκάφους με ε, πάνω από 100 θύματα. Αλλά Ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει κανένα τεστ που να μας επιτρέπει να πούμε με απόλυτη, ασφα... με απόλυτη βεβαιότητα ότι το αεροσκάφος είναι ασφαλές. Κάνετε τους ε, ίδιους ελέγχους πάντα δεν το νομίζω. Εμείς ανταποκριθήκαμε στα αιτήματά σας. Αυξήσαμε τα κονδύλια που διαθέτετε. Αυξήσαμε το προσωπικό που ζητήσατε. Τώρα πρέπει εσείς να ανταποκριθείτε και να κάνετε καλή δουλειά. Με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζονται ορισμένα πράγματα. και το να μην αντιμετωπίζονται σωστά τα πράγματα δεν είναι μια ικανοποιητική κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο, θα, τον λάβω εγώ. Κύριε Κούντου, καταρχήν θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπαν κι άλλοι ως προς τις πιστοποίησεις τρίτων χωρών, την αδειοδότηση για τρίτες χώρες. Το βρεθούμε στη δεύτερη θέση στην εκλογική μου περιφέρεια στο, στην Αγγλία ε, βλέπω ότι μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Μιλάμε για την ευημερία των ζώων. Πρέπει να σώσουμε τις φάλενες και ούτω καθεξής. Αλλά έχουμε πιλότους οι οποίοι πραγματικά μένονται κατά των τρίτων χωρών, κατά τρίτων χωρών και ως προς την πιστοποίηση IMC, τη βαθμολόγηση IMC, γιατί θα χρειαστεί ε, ένα full instrument, full instrument rating 20.000 ευρώ. Βεβαίως το θέμα δεν αφορά ε, μόνο τα ιδιωτικά αεροσκάφη που πέφτουν από τους Ιρανούς, αλλά βεβαίως υπάρχουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη αναψυχής. Για να δούμε μόνο αυτούς. Δείτε τη βαθμολόγηση IMC του Ηνωμένου Βασιλείου και τις περικοπές της αδειοδοτήσεις ε, τρίτων χωρών. Έχω και άλλα σημεία. Ένα ίσονος σημασίας και ένα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν υποχρεωτικοί ε, ε, νόμοι που αφορούν τους αεροδιαδρόμους γιατί εκεί που υπάρχουν υπερβάσεις των αεροδιαδρόμων τα αεροπλάνα σταματούν εκτός και αντίθετα έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα κενό μετά από τον αεροδιάδρομο και μετά να υπάρχει, παραδείγματο χάρη, ένας γκρεμό ή ε, μία περιοχή που να αφορά σιδηροδρόμους. Να προσκρούει κανείς σε μία ζώνη με σιδηροδρόμους. Στη ΣΥΠΑ η συγκυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης, δεν πρέπει να έχει πιστοποιηθεί επί του αεροσκάφους το οποίο οδηγεί. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες συνειδητοποιούν ότι όταν πετάξουν στις ΗΠΑ μπορεί να έχουν στο πιλοτήριο ένα μέλος το οποίο δεν έχει πιστοποιηθεί για το αεροσκάφος που οδηγεί. Ίσως αυτό είναι ένα ζήτημα για τις ΕΠΑ, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς έτσι ώστε στο πιλωτήριο να υπάρχει πλήρης πιστοποίηση και από τα δύο μέλη όταν πετά το αεροσκάφος στην Ευρώπη. Τι διαδικασίες υπάρχουν για να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Η κυρία Φώστερ μίλησε για το εξή, για τα EU Ops. Εγώ πέρασα από το καθαρτήριο του Δάντι έτσι ώστε να έχουμε σωστά EU Ops. Αλλά αυτό δεν αναφέρθηκε καν από την Επιτροπή γιατί φαινόταν δύσκολο θέμα. Άρα με ενοχλεί το ζήτημα. Όταν ε, ακούω για ε, διπλασιασμό χωρίς να επανέλθει κανείς στο κοινοβούλιο, διότι οποιοδήποτε τροποποίηση στα όψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτογενής νομοθεσία και θα πρέπει να αναπαιχθεί σε αυτή την Επιτροπή. Γιατί είχαμε επιδείξεις, έχουμε πολλές αεροεπιδείξεις με πολλά ατυχήματα. Και πολλές φορές υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους οι πιλότοι. Και με ανησυχεί το ζήτημα. Δηλαδή φαίνεται ότι ακούτε περισσότερο τους πιλότους και όχι τις αεροπορικές εταιρείες. Βεβαίως πρέπει να ακούτε τους πιλότους αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες. και τη στιγμή που οι πιλότες λένε ότι τα OPS της Ευρωπαϊκής Ένωσης σοκάρουν και θα πρέπει να ακολουθήσουμε το σύστημα των ΙΠΑ, το αντίστροφο μου λένε οι ΙΠΑ. Δηλαδή ισχύει αυτό και το αντίστροφο. Γίνονται συνεχείς μελέτες και εκτιμήσεις, αλλά θεωρούν οι αεροπορικές εταιρείες ότι δεν εισακούονται όπως είπε και η κυρία Φώστερ, δηλαδή εισακούνται μόνο τα συνδικάτα των πιλότων. Εδώ δεν πρόκειται για μια επιτροπή κοινωνικού διαλόγου. Θα πρέπει να διαβουλεύεστε με τους πάντες. Εγώ προσπάθησα να φτάσουμε σε μια συμφωνία για τις ώρες πτήσης και δεν το θέλαν ίδια οι πιλότοι. Τα άλλα συνδικάτα το ήθελαν, όχι οι πιλότοι όμως. Και δεν θα ήθελα να τα έχουμε δει όλα αυτά εν λεπτομερία. Και παράλληλα τα όψ να μην ακολουθούνται. Δηλαδή η Αυστρία δεν είχε περιορισμό χρόνου πτήσης. Δεν μπορούμε να υποσκαπτόμαστε χωρίς να έχουμε τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να το καταστήσω απόλυτα σαφές. Μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι σε οποιαδήποτε συζήτηση για τα όψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακούσετε τους πάντες από όλο το φάσμα της βιομηχανίας. Και αυτό το ερώτημα το υποβάλλω και στην Επιτροπή. Είσαστε διατεθειμένη να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία μέχρι το τέλος, γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε μια πραγματική συζήτηση. Λυπάμαι που επιμένω, αλλά πια βαρέθηκα. Βαρέθηκα να υποσκάπτονται τα ΟΠΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το καλύτερο σύστημα που έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ. Κύριε Γκουντού. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αρχίζοντας με τη δικό σας βασικό ερώτημα, κύριε Σίμψον. Θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε. Ο κανονισμός μας επέβαλε να ξαναδούμε το θέμα. Δεν τον έφτιαξα εγώ τον κανονισμό, αλλά αναφέρεται στον κανονισμό ότι πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Και αυτό κάνουμε. Διότι το γράψατε εσείς, το, προ... το... εσείς τον κανονισμό. Μας λέτε ότι ακούμε μόνο τους πιλότους. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας ισορροπημένη, ισορροπημένη διότι συμμετέχουν σε αυτήν πέντε ε, ε, οργανισμοί, πέντε αεροπορικές εταιρείες και πέντε εκπρόσωποι των πιλότων. Συν ο οργανισμός, η ΆΣΑ, υπό την προεδρία κάποιου ο οποίος αναγνωρίστηκε από τις αεροπορικές εταιρείες είναι ο κύριος Βόλς, ο κύριος Σπινέτα, ο κύριος Μαϊρούμπερ, σαν κάποιος, έτσι τον αναγνώρισαν, τον παραδέχθηκαν, ότι είναι απόλυτα ικανό άτομο και απόλυτα κατάλληλο για να προεδρεύσει αυτή τη ομάδα. Και το ίδιο ισχύει για τους πιλότες. πιλότους. Πρόκειται για τον κύριο Κότσεν της Επιτροπής. Υπό την προεδρία του κυρίου Κλοντσέν, λοιπόν, αυτή η ομάδα εργασίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, ασχολείται με την τροπολογία των κανονισμών. Δεν ξέρω πια σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει, θα τα έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου και θα δούμε τότε όταν θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά του πού βρισκόμαστε και βεβαίως θα εμπλακίσει όλη αυτή τη διαδικασία το Κοινοβούλιο διότι θα έχει λόγο για τα όψ και ειδικότερα για αυτά τα πακιού. Δεν λοιπόν μπορώ να δεχθώ αυτό που μα είπατε ότι ακούμε μόνο του πιλότους, ότι επισκέφθηκε όλες τι αεροπορικέ εταιρείες, της ενώση πιλότων και ο κύριο Κλωτσέν εργάζεται σε μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα ισορροπημένη ω προ την κατανομή των μελών τη. Συμφωνείτε? Εγώ σα λέω ότι μα λένε εμά. Και δεν είναι αυτή η απάντηση που έχουμε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το παρελθόν αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ξαναδείτε την ΕΑΣΑ. Δεν, δεν σας λέμε να ξαναδείτε, να αναθεωρήσετε την ΕΑΣΑ. Δεν θέλουμε να αλλάξετε οτιδήποτε, διότι αν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, αυτή την αλλαγή πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή σας. Και για αυτό το θέμα, ο κύριος Σεν έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να έχουμε ένα ενιαίο σαπακιού και για τις αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούσαμε να έχουμε κάτι διαφορετικό για, για, για τις διάφορες κατηγορίες αεροσκαφών, αλλά εφόσον πρόκειται για πολιτική απόφαση, την ευθύνη θα την αναλάβει εκείνος και για το ΣΑΠΑΡΚΙΟΥ θα μας δώσει εκείνος συμπεράσματα. Αλλά διαπιστώνω ότι κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το έργο της ΕΑΣΑ που θέλω να τις διορθώσω. Προσπάθησα να το κάνω για το Fees and Charges Θέλω τώρα να διορθώσω τις φήμες που κυκλοφορούν για την ε, ε, όλη διοίκηση της ΕΑΣΑ ε, και της αεροπορίας. Εδώ και πέντε χρόνια, εδώ και πέντε χρόνια με τις ενώσεις τις εκπροσωπευτικές ενώσεις της Γενικής Αεροπορίας έχουμε κάνει δουλειά, έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο δράσης που το επεξεργαστήκαμε μαζί τους για την πιστοποίηση, για, για την συντήρηση των ελαφρών αεροσκαφών Υπάρχει ήδη μια τροπολογία που έγινε δεκτή, που ισχύει πλέον, τις άδειε των πιλότων και προτείναμε στον κανονισμό FCL ένα basic label για τη γενική αεροπορία, για την ε, αεροπορία ε, αναψυχής. Αυτός ο κανονισμός βρίσκεται στο τραπέζι της Επιτροπής στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας. Δεν μπορείτε να μας πείτε ότι δεν δέχομαστε αυτά που προτείνει η Γενική Αεροπορία, διότι αυτό ακριβώς μας είχαν ζητήσει οι εκπρόσωποι της Γενικής Αεροπορίας. Προτείνουμε μια απλουστευμένη άδεια, μια απλουστευμένη ιατρική εξέταση, μια πιστοποίηση των ε, απλουστευμένη διαδικασία πιστοποίησης. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε φήμες, αλλά πάνω σε γεγονότα αυτό που σας προσκομίζω σήμερα είναι γεγονότα. Αυτά κάναμε και στην γνωμοδότηση που υποβλήθηκε για το FCL στην Επιτροπή θα βρείτε το Basic Lappel. το basic, ε, τα, τα βασικά, τις βασικές απαιτήσει για τους εξεταστές κλπ. ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα της Γενικής Αεροπορίας, τα κάναμε. Κύριε Γκουντού, κάποιος πρέπει να μας δώσει κάτι. Όλες αυτές οι επιστολές που λάβαμε ε, θα μπορούσα να απαντήσω λέγοντας ότι ο κύριος Γκουντού θα απαντήσει σε αυτές όλες τις επιστολές και θα τους προτείνω να τις στείλουν σε εσά και εμείς θα απαντήσουμε. Αυτός ο κανονισμός θα μπει στη διαδικασία της επιτροπολογίας και του Κοινοβουλίου. Ξέρω τι προτείναμε, δεν ξέρω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, η έκβαση του κανονισμού. Ε, το, η βαθμολογία AMC. Είμαι ο πρώτος που λέω ότι εάν πιλότ, ένας πιλότος βρεθεί σε μία δύσκολη θέση διότι για έναν απροσδιόριστο λόγο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δηλαδή, ε, ακραίες καιρικέ συνθήκες. Ε, εάν είχε κατάρτιση IMC, τότε θα τα καταφέρει, μάλλον θα τα καταφέρει, έχει περισσότερες πιθανότητες. Αυτό το έχουμε πει αρκετές φορές σε σχέση με το, τη βαθμολόγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη πλαισίωση γιατί έτσι ε, βελτιώνεται η ασφάλεια. Δηλαδή ένα ρυθμισμένο πλαίσιο μέσα στα πλαίσια της βαθμολόγησης AMC του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι όμως η μόνη χώρα όμως που δέχεται αυτή τη βαθμολόγηση IMC. Όταν όμως ένας πλότος βρίσκεται πολύ κοντά στα σύννεφα και πρέπει να βγει, εάν έχει κατάρτιση IMC, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρει με επάρκεια. Άρα είμαστε υπέρ της βαθμολογίας IMC, με τη σωστή ρύθμιση και πλαισίωση. J'en viens aux, Ως προς τις ε, πιστοποίησεις τρίτων χωρών στο FCL, προτείνουμε αυτό που συμβαδίζει με τις οδηγίες σας. Αυτό είχατε ζητήσει από το βασικό κανονισμό. Απλώς είπαμε ότι ένας πιλότος που πετάει στην Ευρώπη πρέπει να έχει ευρωπαϊκή άδεια. Προτείναμε ένα σύστημα μετατροπής γρήγορα και εύκολα των ξένων αδειών σε ευρωπαϊκές. Εάν πρόκειται για αμερικανικές άδειες, εάν ε, επέλθει συμφωνία, διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ, αυτό θα βοηθήσει αυτή τη μεταφορά και αποδοχή των αμερικανικών αδειών στην Ευρώπη. Κάνουμε ακριβώς αυτό που μας ζητήσατε. Οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να δώσουν κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι αν οι, οι ΗΠΑ αρνηθούν την αμοιβαία αναγνώριση, πιέζεται τους δικούς μας πιλότους να κάνουν ένα τεστ ευρωπαϊκό και το κόστος ε, αυτού δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπό... υπόψη. Αν αφαιρέσουμε το θέμα της αμερικανικής συνεργασίας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν, είναι ότι θέλουμε ε, ή δεν θέλουμε ευρωπαϊκή άδεια, είναι το κόστος μιας ευρωπαϊκής άδειας. Κύριος Γκουντού, μπορώ να σας πω απλώς ότι υπάρχει ο βασικός κανονισμός σχετικά με την ευρωπαϊκή άδεια και προτείναμε μια εύκολη μετατροπή αμερικανικών ή άλλων αδειών σε ευρωπαϊκή άδεια. Όντως με ένα μικρό τεστ, απλώς ε, για να αποδειχθεί ότι ο εν λόγω πιλότος γνωρίζει τους επιχειρησιακούς κανόνες και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο που είναι πολύ διαφορετικός από τον αμερικανικό εναέριο χώρο. Πλήρωμα καμπίνας και ιατρικό ενδεχομένως πλήρωμα. Διαβάζω το παράρτημα όπου ξεκάθαρα λέει ότι το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να έχει μία βεβαίωση και τη βεβαίωση αυτή πρέπει να την έχει το πλήρωμα καμπίνας όσον αφορά και τεχνικά θέματα που θα αποδεικνύει, δηλαδή ότι έχουν την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και δεύτερον και μία βεβαίωση για τα ιατρικά θέματα με βάση την βέλτιστη ιατρική πρακτική. Αυτά λέει ο βασικός κανονισμός στο παράρτημα. Προσπαθήσαμε στην πρόταση που έγινε Προσπαθήσαμε, τηρώντας αυτά τα οποία υπάρχουν στο βασικό κανονισμό, να εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα όσον αφορά την ιατρική εξέταση. Δεν έγινε αποδεκτό από τα κράτη-μέλη στην επιτροπολογία και εδώ αντιμετωπίζουμε μείζωνα δυσκολία. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θέλουν ε, κάτι που θα ανταποκρίνεται στο ότι ο καθένας θα κάνει τα δικά του. Πού είναι η ομοιομορφία και ε, οι ίσοι κανόνες ανταγωνισμού που ζητά η Ευρώπη. Βρισκόμαστε στο στάδιο υποβολής προτάσεων τώρα και ε, η γενική κατεύθυνση είναι μια μείωση των απαιτήσεων όπου αυτό είναι δυνατόν. Όμως πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν στο βασικό κανονισμό μια ιατρική βεβαίωση που βασίζεται στις βέλτιστες ιατρικές πρακτικές. Όμως τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή στη διαδικασία της Επιτροπολογίας θα πρέπει να δώσουν την τελική του μορφή στο κείμενο. Εμείς απλώς υποβάλλουμε προτάσεις. Να σας δώσω το λόγο, αλλά μην ε, καθυστερήσετε παρακαλώ. Ε, κοιτάξτε, ο κύριος Γκουντού ε, μας έκανε τα σχόλιά του. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε κάτι. Και αν δείτε το θέμα των ιατρικών βεβαιώσεων, κάπου λέμε για μία φορά κάθε έξι μήνες. Το κόστος για κάτι τέτοιο θα είναι τεράστιο. Και οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες κάνουν ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό όταν αρχίζουν, την, ε, όταν προσλαμβάνονται, αλλά όχι αργότερα. Και ε, εσείς ως οργανισμός ασφάλειας, ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει από το Κοινοβούλιο, εσείς θα λάβετε από τα θεσμικά όργανα διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε. Αν δεν είναι καθαρά θέματα ασφαλείας, γιατί αυτό δεν είναι θέμα ασφαλείας καθόλου θα πρέπει να είστε σε θέση να πείτε, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα θέμα που είναι θέμα ασφαλείας, πρέπει να επανέλθουμε και να το συζητήσουμε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Εσείς ως ΕΑΣΑ πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να ξέρετε ότι όταν σας στέλνουμε κάποια νομοθετικά κείμενα έχετε τη δυνατότητα να επανέλθετε και να πείτε ότι πρέπει να το συζητήσουμε και να μας πείτε ότι δεν θα δουλέψει στην πράξη ή δεν θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε όσο εύκολα θα θέλαμε για τον α ή β λόγο. Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Φώστερ, πουθενά στην πρόταση που κάναμε δεν θα δείτε ανάγκη να γίνεται ιατρικός έλεγχος κάθε έξι μήνες πουθενά. Εγώ σέβομαι τη γνώμη του λαού, σκέπτομαι, ε, σέβομαι τη γνώμη του Κοινοβουλίου και όταν μου ζητάει το Κοινοβούλιο να κάνω κάτι, το κάνω. Κάποια σημεία τώρα που αφορούν άλλα θέματα, διότι νομίζω ότι καλύψαμε το FTL και το FCL λίγο πολύ. Το Airbus το πρόβλημα του κινητήρα. νέος κανονισμός για το Airbus 380 και για τα τυχήματα. διότι αυτός ο κανονισμός, αυτές οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ένα ρόλο για τον, την, τον οργανισμό. Ο προηγούμενος κανονισμός είχε θεσπιστεί πριν από την ίδρυση του, της ΑΣΑ, οπότε δεν, μπορεί, δεν είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην εκπόνηση αυτών των νέων ρυθμίσεων. Τώρα έχουμε αναλάβει σύμφωνα, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό το ρόλο του Συμβούλου και χάρη σε αυτό θα έχουμε πρόσβαση εφόσον υπάρχει ανάγκη και το ταχύτερο δυνατό στα δεδομένα ασφάλειας τα οποία χρειαζόμαστε εμείς για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Η δουλειά μας συνίσταται στο να ε, βλέπουμε, να εξετάζουμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα άμεσης, άμεσης βελτίωσης της ασφάλειας των αεροσκαφών και να μην περιμένουμε συμπεράσματα μετά από ατυχήματα για να το κάνουμε αυτό. Αν έχουμε τη βεβαιότητα ότι ε, αναλαμβάνοντας δράση πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας ε, θα είναι σημαντικό. Ο κανονισμός αυτός μας δίνει πρόσβαση σε μία δεδομένων, ναι. τουλάχιστον σε ορισμένα άτομα και κανονίο, κατανοώ ότι αυτό γίνεται για λόγους εμπιστευτικού χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση για λόγους απορρίτου. Αυτό ζητούσαμε εδώ και πολύ χρόνο, διότι οι πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε με βάση την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Έκερς δεν θα είχε κανένα νόημα για τους αναλυτές μας. Χαίρομαι λοιπόν που εισήχθη αυτός ο νέος κανονισμός και ελπίζω να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Ως προς το ατύχημα της Κουάντας του Airbus 380, ε, πρόκειτο για ένα πρόβλημα στον κινητήρα, γιατί ο κινητήρας είναι της Rolls-Royce. Η έρευνα διενεργείται τώρα, δεν έχει λήξει η αποσυναρμολόγηση του κινητήρα, άρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σήμερα. Αυτό που είναι σαφές είναι το εξής για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό τον κινητήρα. Μόνο η Qantas βρήκε κάποιο πρόβλημα στους κινητήρες. Singapore Airlines ξαναείδε όλους τους κινητήρες, δεν βρήκε καμία δυναμία. Δεν βρήκε κανένα κρίσιμο σημείο. αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οδό που πρέπει να διερευνήσουμε για να ανακαλύψουμε και να διαπιστώσουμε τα αίτια αυτού του ατυχήματος. ο εκπρόσωπος της Κουάντας ε, μας είπε άλλα πράγματα στο Λονδίνο, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ε, το τι προκάλεσε το ατύχημα, ε, γιατί δεν το ξέρουμε. Σχόλια εκτός μικροφώνου. We know, το μόνο που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε είναι το εξής, λέει ο πρόεδρος και διακόπτη. Όπως σας είπα στην προηγούμενη συζήτηση, χρησιμοποιούμε τον όρο ατύχημα. Δεν ήταν ένα ατυχές συμβάν, ένα συμβάν δεν ήταν ατύχημα στην Qantas. Κάθε αεροπορική εταιρεία έλεγξε τους κινητήρες της και η Κουάντας δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Αλλά δεν πρέπει να φτάνουμε σε γρήγορα ε, από, ε, συμπεράσματα για το τι δημιούργησε το ατύχημα μέχρι ότου έχουμε την ε, πλήρη, τα, τα πλήρη συμπεράσματα από την έκθεση. Συμφωνώ απολύτως και όντως δεν μπορούμε να λάβουμε θέση μέχρι ότου καθοριστούν οι αιτίε του συμβάντο. Όσον αφορά την κρίση με την έκρηξη του ηφαιστείου, ο οργανισμός μας ε, συμμετέσχει σε διάφορες δράσεις όσον αφορά την ε, αξιοπλοεία και ε, ταχαίω συνεργαστήκαμε με τους κατασκευαστές κινητήρων για να ξέρουμε τα όρια αυτών των κινητήρων ένα πολύ δύσκολο έργο και παραμένει πολύ δύσκολο το έργο αυτό. Οι κατασκευαστές των κινητήρων ε, δεν μπορούν να δεσμευθούν για την ποσότητα στάχτης που μπορεί να εισροφήσει ένας κινητήρας μέχρι ότου φτάσει σε πρόβλημα και τι πρόβλημα θα είναι αυτό. Θα είναι πρόβλημα συντήρησης ή σοβαρότερο πρόβλημα. Εργαζόμαστε λοιπόν σε συνεργασία με τους κατασκευαστές και στο πλαίσιο της ε, ΙΚΑΟ και αν ε, κάτι πρέπει να καθοριστεί, θα καθοριστεί σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι τεράστια η δυσκολία, διότι κάθε ηφαίστειο έχει διαφορετικό τύπο στάχτης, διαφορετική σύνθεση της στάχτης και η πυκνότητα της στάχτης δεν είναι η ίδια. Είναι δύο οι κατευθύνσεις πάνω στις οποίες δουλεύουμε. Καταρχήν αντίσταση των κινητήρων στη στάχτη, αλλά και πυκνότητα στάχτης στην ατμόσφαιρα. Και έχουν πολλή δουλειά και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες για να ποσοτικοποιήσουν την ποσότητα στάχτης που διαχύθηκε τελικά στην ατμόσφαιρα και που μπορεί να ισροφηθεί από τους κινητήρες αεροσκαφών συντονίζουμε τις δραστηριότητες των κατασκευαστών μαζί με τον ΙΚΑΟ, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και προσπαθούμε να συντονίσουμε και τα μέτρα, ε, να δούμε δηλαδή τους, ε, ποιοι είναι οι οργανισμοί που μπορούν ε, να κάνουν τέτοιες μετρήσεις στάχτης και πυκνότητας. Πολύ δύσκολα έργα όλα αυτά που προσπαθούμε να τα διεκπαιρεώσουμε με επιτυχία. Κλείνοντας, θα μιλήσω για το θέμα των τελών και εισφορών. Γιατί προτείνεται ένα καινούριο σύστημα. Μα επέπληξαν διότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικέ οι τιμέ. Ορισμένε δραστηριότητε αμείβονταν πάρα πολύ ακριβά, τα πιστοποιητικά τύπου παραδείγματο χάρη, ενώ άλλε δραστηριότητε δεν αμείβονταν επαρκώ όπως παραδείγματο χάρη για την παρακολούθηση τη αξιοπλοεία. Δουλέψαμε λοιπόν με κάποιο σύμβουλο επιχειρήσεων και με μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κλάδος, ε, διάφοροι φορείς, ε, μια ευρεία ομάδα εργασίας για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε νέες τιμές που θα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του κόστους και πάλι αφήσαμε κατά μέρο του μικρού κατασκευαστέ, ώστε να μην φύγονται κατά κανένα τρόπο και να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο κόστο που επιβάλλεται στου μικρού κατασκευαστέ. Αυτό κάναμε λοιπόν και τώρα θα έχουμε τις νέες τιμές ε, για τις νέες δραστηριότητες ε, που δεν είναι πολλές, δεν θα είναι πολλές αυτές οι τιμές Υπάρχει το θέμα, παραδείγματο χάρη, της ε, εποπτείας των ευρωπαϊκών ε, προμηθευτών για το ATM. Θα πρέπει να δούμε κάποιους προσωμιωτέ πτήσει. τέτοιου είδου θέματα. Ξέρετε για την, αρμοδιότητα, για την επέκταση τη αρμοδιότητας ε, του οργανισμού είχαμε μικρό πεδίο δραστηριοτήτων και τα κράτη-μέλη κράτησαν το μεγαλύτερο κομμάτι. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που αφορούν τα κράτη-μέλη, που είναι η τυποποίηση, η έλεγχη στα κράτη-μέλη για να επαληθεύσουμε ότι όντως ε, συμμορφούνται προς τον κανονισμό και ε, οι αναλύσεις τις οποίες επομίζεται το ευρωπαϊκό ε, επίπεδο και εδώ θέλουμε να έχουμε την συνεισφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Για τα δύο σημεία που θέσατε εσείς, ε, για τους διαδρόμους ε, και για τις άδειε πιλότων της ΗΠΑ, θα σας στείλω γραπτός απάντηση. Στην Ευρώπη θέλουμε οι πιλότοι να έχουν, ε, οι συμπιλότοι, οι συγκυβερνήτες να έχουν ε, ίδια πιστοποιητικά τύπου, όπως και οι κυβερνήτες. Δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνηση του αεροσκάφου. Μπορεί να βρεθεί μόνος του ο συγκυβερνήτης και να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, ο κύριος Σίμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Δεν θέλω να απαντήσω σε όλα τα θέματα που ακούσαμε κατά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Πιστεύω και η Επιτροπή πιστεύει ότι το έργο το οποίο κάνει η ΕΣΑ το όψι είναι το πιο επίμαχο θέμα και γι' αυτό αναφέρομαι συγκεκριμένα ε, στο όψι, αλλά όλο το έργο του ΕΑΣΑ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επιμείνω για το όψι για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς πρέπει να λειτουργεί το σύστημα σύμφωνα με τους νομοθέτες. Πρώτο σημείο. Η ΕΑΣΑ ως οργανισμός που προετοιμάζει τα νομοθετικά κείμενα, έχει ένα σημαντικό έργο και σύμφωνα με το βασικό κανονισμό πρέπει να βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία της ε, απαραίτητης νομοθεσίας και βοηθά τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτό είναι το έργο της ΕΑΣΑ. και με τις ε, επεκτάσεις αρμοδιοτήτων Η Επιτροπή παρακολουθεί αυτό το έργο από την αρχή μέχρι τη γνωμοδότηση που δίδει η ΕΑΣΑ και με ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Η ΕΑΣΑ έχει ένα σύστημα διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη και με τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και ιδιαίτερα εκτενές και πολλές φορές έχω αναρωτηθεί μήπως η πολυπλοκότητα αυτού του συστήματος ε, είναι ο λόγος ε, για κάποιες ε, ανησυχίες ή διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στο τέλος, αλλά είναι προσωπική μου ανησυχία αυτή και δεν θέλω να το βάλω αυτό τώρα στη συζήτηση. Όταν εκδώσει την γνωμοδότησή της η ΕΑΣΑ μετά από μακροχρόνια προπερασκευαστική εργασία, η γνωμοδότηση αυτή πηγαίνει στην αρμόδια κανονιστική επιτροπή για να το σκεφτούν και τα κράτη-μέλη και μετά φτάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επομένως, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει μειωθεί καθόλου. Είναι απολύτως τμήμα του συστήματος. Το σύστημα είναι πολύπλοκο, ίσως πιο πολύπλοκο από ό,τι σε άλλους νομοθετικούς τομείς, αλλά υπάρχουν ε, και λόγοι για την πολυπλοκότητα του συστήματος και κυρίως είναι ότι είναι πολύ τεχνικό αυτό το έργο και υπάρχουν και τα θέματα ασφάλειας που χρειάζονται πάρα πολύ καλή προετοιμασία και πυρογνωμοσύνη σε τεχνικά θέματα. Μπορεί να ρωτήσετε τώρα την Επιτροπή ποια είναι η δική μας συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας νομικών κειμένων. Συνεργαζόμαστε με την ΕΑΣΑ και κατά όλη αυτή τη διαδικασία εμείς πάντοτε λέμε στην ΕΑΣΑ τους κανόνες τους οποίους προτείνεται να προσπαθεί να τους αντλείται από υφιστάμενους κανόνες και από το EU OPS, εκτός αν υπάρχει κάποιος απαραίτητος λόγος ασφαλείας κάτι που απαιτεί μια τροποποίηση των ε, όσων ήδη ισχύουν. Και πρέπει να πείτε σε όλους αυτούς που σας κατακλείζουν με emails ποια είναι η αξιολόγηση ασφαλείας σας σε σχέση με τη γνωμοδότηση που έχει εκδώσει η ΕΑΣΑ για την συγκεκριμένη πρόταση. Μπορεί κάποια φορά να υπάρχει κάποιο ζήτημα, αλλά από τη συζήτηση αυτή που ακούσαμε εδώ, νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό που μας είπε η κυρία Φώστερ, παραδείγματο χάρη, ή και άλλοι ομιλητές, το επιβεβαιώνουν. Πιλότες ιδιώτες. Πιλότοι, συγγνώμη, ιδιώτες. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός για αυτά τα θέματα. Και αν θέλουμε να το αναπτύξουμε θα είναι κάτι καινούριο. Και υπάρχει και άλλος τομέας, οι άδειε τρίτων χωρών. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός για το πώς πρέπει να χειριστούμε τις άδειες πιλότων τρίτων χωρών. Και είναι φυσιολογικό ότι η ΕΑΔΣΑ θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ή να μην γίνονται αποδεκτές αυτές οι άδειε. Εκτός αν βρούμε ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα, μια συμφωνία ασφαλείας με την εν χώρα για την αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό θα διευκόλυνε κατά πολύ το έργο μας για την αναγνώριση αδειών τρίτων χωρών. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και πάντοτε, στη συνεργασία μας με την ΕΑΣΑ, αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους υφιστάμενους κανόνες και όταν υπάρχουν κανόνες θα πρέπει να τους λαμβάνουν υπόψη και πάνω σε αυτούς να βασίζονται, εκτός αν υπάρχει κάποιο επιχείρημα περί της ασφαλείας. Όμως, όπως ε, είπαμε, υπάρχουν κάποιοι τομείς και πολλοί από αυτούς τους τομείς έχουν οδηγήσει σε αντιδράσεις από τους ενδιαφερομένους, όπου η ΑΣΑ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία να υποβάλει προτάσεις και εμείς πρέπει να τις επαληθεύσουμε. Τώρα, για το επόμενο σημείο, για το ATM, δεν ήταν τόσο αντιφατικό αυτό το σημείο. Νομίζω ότι εδώ έχουμε καταλήξει σε ένα αποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΑΣΑ, Επιτροπής και Eurocontrol. Και εδώ πάλι Θέλουμε να αντλήσουμε από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και να μην προσπαθήσουμε να εφεύρουμε τίποτα νέο. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία που πρέπει να έχουμε κατά νου. Όταν έρχονται οι προτάσει και πρέπει να τι εξετάσουμε, αυτή είναι η βασική μα αρχή. Ακόμη θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε τομείς όπου δεν υπάρχει εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση υπάρχουν πολύ διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη και θα μπορούσα να σας αναφέρω παραδείγματα. Το, οι άδειε για τους ιδιώτες πιλότους, ε, το Basic Apple μεταξύ άλλων, που είναι ένας τεχνικός όρος. Υπάρχουν πολλές απόψεις ε, των κρατών μελών που δίστανται. Και μέλη της Επιτροπής σας, ε, που άκουσα σήμερα το απόγευμα, εξέφρασαν απόψεις που είναι αρκετά διαφορετικές από τις απόψεις των κρατών μελών με βάση την εμπειρία τους, με βάση του πώς χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος τους, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές στο Βέλγιο, στη Γαλλία κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μια σωστή αξιολόγηση αυτών τα οποία βρίσκονται επιτάπητος και θα ήθελα να σας ε, τονίσω ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν ως διατάξεις πρέπει να ε, αποτελέσουν τη βάση μας πάνω στην οποία θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά τα τέλη και εισφορές, προσπάθησε ο κύριος ε, Κουντού να εξηγήσει το θέμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε ένα κανονισμό τελών και εισφορών στο σύστημα ασφαλείας μας και τώρα. Και γιατί ξεκίνησε κάποια δουλειά αναθεώρησης αυτού του συστήματος. Υπάρχει ένας τυπικός λόγος. Η εντολή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τροποποιούμενο ρόλο. Και αφού έχει αλλάξει ο ρόλος, πρέπει κάπως να ε, αντανακλάται αυτό και στα τέλη και εισφορές που υπάρχουν. Όπως είπε ο κ. Γκουντού, το θέμα που υπευλήθη και στην ΕΑΣΑ και στην Επιτροπή είναι ότι ενδεχομένω θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να αντικατοπτρίζει περισσότερο το κόστος σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα. Και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, θα γνωρίζουν ότι οι συμφωνίες ασφάλειας αεροπορίας που συνάπτουμε με τρίτες χώρες, ήδη έχουμε δύο-τρεις συμφωνίες με τη Βραζιλία και με τον Καναδά, και είναι τεχνικά έτοιμη η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζουμε ότι σύντομα θα προχωρήσει. Μετά από τις συμφωνίες αυτές, ε, η συνέπεια είναι ότι χρειάζεται ένα σύστημα εισφορών και τελών ε, που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος. Και αυτό αποτελεί επαρκή λόγο για να αναθεωρήσουμε το όλο σύστημα, ώστε τελικά να έχουμε μια περισσότερο συνεκτική πρόταση. Η Επιτροπή έχει πλέον ε, τον ε, ρόλο του να προχωρήσει, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκουντού. Αλλά υποφελούμε τις ευκαιρία για να πω ότι όταν αλλάζει κάτι τα τέλη και εισφορές, κανείς ε, δεν μπορεί να τους ικανοποιεί όλους. Θέλουμε λοιπόν πρώτα να λάβουμε υπόψη μας τους βασικούς στόχους, το κόστος θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις εισφορές και στα τέλη. Και όπως ξέρουμε έχουν εξελιχθεί οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΑ και αυτό απαιτεί τροποποίηση του κανονισμού για τα τέλη και εισφορές. Και δεν μπορώ να σας πω σήμερα πριν γίνει η πλήρη συζήτηση με τους πολιτικά ηθήνοντες, ε, τι θα προταθεί. Δεν ξέρουμε τι απαιτείται. Αν θα αλλάξει η γενική διάρθρωση ή όχι. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολύ μικρών φορέων των πολύ μικρών εταιριών, αλλά σίγουρα πάντα θα υπάρχει ε, κάποιος δυσαρεστημένος που θα θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να πληρώνει τόσα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με το κόστος και θέλουμε να μπορούμε να το αποδείξουμε. Κυρία Λίχτενπέργκερ. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα που έχει σχέση ε, με κάτι που δεν απαντήθηκε ε, από όσα άκουσα. Στο θέμα των πιλότων και του χρόνου ανάπαυσης, πάντοτε η Επιτροπή και η ΕΑΣΑ μας έλεγε ότι θα γίνει μια μελέτη σχετικά με την κόπωση και δεν την έχω δει αυτή τη μελέτη. Υπάρχει τέτοια μελέτη και αν υπάρχει θα μας τη δώσετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει άμεση σχέση με αυτά τα οποία συζητήσαμε. Και το αν θα πρέπει να υπάρχουν ιατρικά δεδομένα, όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά γενικά. Έτσι είχαμε ξεκινήσει όταν το προτείναμε. Ε, και αν δεν υπάρχει τέτοια μελέτη, γιατί μας την είχατε υποσχεθεί. Και θα ήθελα να πω ακόμη ότι δεν συμφωνούμε όλοι με την άποψη ότι πρέπει να εγκρίνουμε τις άδειες πιλότων από άλλες χώρες. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω σε σχέση με τις άδειες από τις ΗΠΑ. Δεν συμφωνούν όλοι. Η μόνη μελέτη που είδαμε ήταν η έκθεση μελούς, η οποία αμφισβητείται. Και ο ίδιος ο συντάξης μου είπε ότι, ο ίδιος ο συντάξης μου είπε ότι δεν είναι επαστημονική η έρευνα. Είναι η μόνη που έχει αναλυφθεί. Yeah, Κανένας δεν θα την υπέγραφε, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είναι η, η μόνη που γνωρίζω. And that's confirmed. That's the only one. Είναι η μοναδική. Please for the future για το μέλλον ε, μην κάνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Η κυρία Μάισνερ θέλει να πείτε. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε η Εύα Λίχτενμπέργκερ. Για τη μελέτη για την κόπωση ήδη απαντήθηκε η ερώτηση. Από ό,τι ξέρω, και από τις ενώσεις των πιλότων. Η χρόνια ανάπαυσης είναι πολύ μικρή και νομίζω ότι αυτό παίζει και άμεσο ρόλο στα θέματα ασφάλειας. Ε, ήταν ένα θέμα του ΠΟΕ σε σχέση με την Boeing έναντι της Airbus. Αλλά από όσο γνωρίζω, όταν ρώτησα κατά πόσο ήταν επιστημονική μελέτη, ο συντάκτης μου είπε ότι όχι. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε ή να ρωτήσετε. Εάν όχι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους. Πολύ ζωηρή συζήτηση και άκρος ενδιαφέρουσα όπως αναμενόταν και ευχαριστούμε κύριε Γκούντου που ήρθατε και μας είπατε πώς έχει η κατάσταση και που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Καταλαβαίνετε τι μας απασχολεί. Ο κύριος Σίμπον είπε πολύ σωστά ότι υπάρχει πρόβλημα στην κατάρτιση κανόνων. Έτσι έχει το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και ευχαριστώ και τους βουλευτές για την εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ και γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστεί ο Πρόεδρος τους ε, Διερμηνείς και θα επανέλθουμε στην τρίτη 30 του μηνός στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ.